I start now. Good morning, everybody. It's not so much everybody, but my two colleagues, thank you for being here. We start with point nine, European Year for... Αρχίζουμε το σημείο 9. Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Δεσυνογό Γύρανσης. Ας μιλήσουν οι πιο νέοι. Χάνω, έχεις το λόγο. Voisi sanoa, että kun την τελευταία φορά που το συζητήσαμε κατά την πρώτη ανάγνωση τότε είχα πιο κοντά μαλλιά και φαινόμουν ακόμα πιο νέος. Τέλος πάντων έχουμε και έξι εξελίξεις αυτές τις εβδομάδες που μεσολάβησαν οπότε έχουμε γίνει σοφότεροι ενδεχομένω και όπως είπαμε την τελευταία φορά όσον αφορά το σχετικό κοινοτικό πρόγραμμα και όσον αφορά το πώς κάποιος μπορεί και να γυράσκει αλλά και να είναι ενεργός είπαμε να τονίσουμε τα θέματα της ε, σωματικής δραστηριότητας, της φυσικής αγωγής σε σχέση με τη γύρενση. Του χρόνου επομένως και το 2012 θα είναι η τότε ενεργού γύρανσης. Και έτσι θα έχουμε επίσης και εθελοντική δραστηριότητα σε σχέση με την ενεργογύρανση. Αυτή η εθελοντική δραστηριότητα θα αναλυφθεί από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Να μην ξεχνούμε ότι όταν κανείς ε, μεγαλώνει γίνεται πιο έμπειρος. Και επίσης αποκτά περισσότερη γνώση η οποία πρέπει να μεταδοθεί στις νεότερες γενιές. Και γι' αυτό θέλω να πείσω την προσοχή σας στο ότι κάποιος όταν μεγαλώνει μπορεί να συμμετέχει σε δραστηριότητε, αλλά και σε πνευματικές και σε σωματικές δραστηριότητες, τόσο ώστε και πλευρά σωματικής αλλά και πνευματικής και ψυχικής ε, να ωφελείται. Επομένως, όταν κάποιος μπορεί ακριβώ να φροντίσει όλες αυτές τις πτυχές της προσωπικότητάς του, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Είναι και επίκαιρο το θέμα σήμερα, μια που όπως γνωρίζετε έχουμε ένα σωρό αρνητικά τα οποία συμβαίνουν όσον αφορά την Ευρώπη. Επίσης ε, θεωρείται ότι τώρα ήρθε η ώρα του να στεξιοδοτηθεί η γενιά του baby boom, όπως λέγεται, αυτής της ε, έκρηξη γεννήσεων και επομένως τώρα αξίζει να αναδείξουμε το ότι τα πρόσωπα δεν είναι ούτε απλή αριθμή, ούτε απλά λιθαράκια στην αύξηση του ΑΕΠ, αλλά είναι κάτι παραπάνω. Και επομένως και κατά την πρεσβύτερη ηλικία η ζωή μπορεί να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα να έχει δραστηριότητες και άρα θα πρέπει να δούμε τι ποιοτικά στοιχεία έχει αυτή η φάση της ζωής, τι είναι τα... ποια, ποια είναι η προστιθέμενη αξία. Να το συζητήσουμε, να ακούσω τις προτάσεις των συναδέλφων. Και ξέρετε, έχουμε και ένα ερωτικό τραγούδι στην Φινλανδία που κάποιος λοιπόν τραγουδά στην ε, αγαπημένη του και ε, ετοιμάζονται να περάσουν λοιπόν τη βραδιά της ζωής τους και τραγουδάει και ε, λέγοντας ε, ναι, ναι, να γεράσεις, να σχημείνεις, αλλά με ένα χαριτωμένο τρόπο. Να, να τι μπορούμε να κάνουμε μένα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν ε, κατάλαβα απόλυτα τα λόγια από το τραγουδάκι το φιλανδικό, αλλά θα ζητήσω από τους συναδέλφους να μου πούνε πώς ε, ονομάζεται, πώς, ε, ε, λέγεστε Ιωάννα είναι ένα πολύ δύσκολο πολωνέζικο όνομα, γι' αυτό εντάξει και Τζοάννα να μην πείτε, μια χαρά είναι. Λοιπόν, να συνεχίσω πρόεδρε. Ευχαριστώ τον συνάδελφο για τις παρατηρήσεις που έκανε επί της γνωμοδοτήσεως. Εγώ από πλευρά ε, ΕΛΚ είμαι σκιώδη ηγήτρια και θα ήθελα να παρουσιάσω τις παρατηρήσεις μου. Ε, ακολουθούμε μια διαδικασία, μάλλον πολύ διαδικασία κατά τη διάρκεια του βίου μας και σε πολλέ ε, φάσεις ε, είμαστε ικανοποιημένοι, δεχόμαστε τις εξελίξεις. Τώρα, η ενεργός γύρανση έχει οριστεί από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στη δεκαετία του 1990 και αφορά την οικονομική, την ε, κοινωνική, την πνευματική, την διανοητική ε, ζωή, φυσικά με την συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, σωματικές ε, δραστηριότητες κλπ. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τον άνθρωπο κατά την γύρανση του ε, στους ηλικιωμένους υπάρχουν ποικίλα επίπεδα υγείας και διάφορα επίπεδα ανεξαρτησίας. Χρειάζεται λοιπόν να αποφασίσουμε αν για να προσδιορίσουμε τους ηλικιωμένους θα προσπίσουμε και κάποιο επιπλέον κριτήριο πέραν το ηλικιακό. Εγώ είμαι υπέρ του εθελοντισμού ως ε, δραστηριότητα για τους ε, ηλικιωμένους. Το... Σε λίγο θα έχουμε το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού για τους ε, ηλικιωμένους και την επόμενη χρονιά προλέπονται δραστηριότητες για την εργογύρανση. Λοιπόν, το ζήτημα αυτό, όπω καταλαβαίνετε, δεν αφορά μόνο τους νέους και την συμπεριφορά αυτών, αλλά θα πρέπει να δημιουργήσουμε ιδιαίτερο ενθουσιασμό για τον ε, εθελοντισμό σε ε, όλα τα επίπεδα. Οι ηλικιωμένοι πρέπει να είναι σε θέση να βελτιώνουν τις γνώσεις τους ε, προκειμένου να διατηρήσουν και να διαβρύνουν τις ψυχικές, σωματικές ικανότητες, σωματικές ικανότητες τους. Στην Πολωνία είναι πολύ γνωστά τα πανεπιστήμια της τρίτης ηλικία. Είναι μια πρωτοβουλία πάρα πολύ σημαντική η οποία χρειάζεται να διευρυνθεί περαιτέρω. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν οι ηλικιωμένοι δυνατότητες επαφής με αυτά τα πανεπιστήμια, με πολιτιστικά κέντρα. Πέραν από τον τομεακών γνώσεων, ε, συνήθως ε, μαθαίνουν ξένες γλώσσες, ε, μαθαίνουν μαγειρική, ε, ηλεκτρονικούς υπολογιστέ, υπάρχουν διάφορα σεμινάρια χορού, υπάρχουν επίσης πολλές βιβλιοθήκες οι οποίες είναι στην διάθεση των ηλικιωμένων προσώπων. Ε, είναι ιδιαίτερα δεδομένα λοιπόν όλα αυτά, αλλά χρειάζονται και κάποια οικονομική στήριξη. Χρειάζεται λοιπόν κατά το έτος της ενεργού γύρανσης ε, να προαγάγουμε αυτές τις ε, δραστηριότητες, αυτές τις πρωτοβουλίες και απαραίτητα είναι και η άθληση για τους ηλικιωμένους προκειμένου να διατηρήσουν την καλή σωματική τους κατάσταση πρέπει να έχουν ε, δυνατότητα πρόσβασης ε, στους ε, αθλητικούς συλλόγους, στα γυμναστήρια κλπ. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε φυσικά και το ζήτημα της γενικότερης υγείας σας. Ευχαριστούμε λοιπόν το 2012 για να προαγάγουμε την δυνατότητα πρόσβασης των ηλικιωμένων σε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Πρέπει να διατηρήσουμε την σωματική και ψυχική υγεία, επαναλαμβάνω. Χρειάζεται λοιπόν συντονισμένη δράση σε περιφερειακό, τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερη προσοχή χρήζουν ε, ε, τα πιο φτωχά στρώματα και αυτό που έχει σημασία είναι να μπορέσουμε να εγγυηθούμε ότι η διαδικασία γύρανσης να συνδέεται με μια ε, καλή υγεία και με συμμετοχή σε πολιτικές ε, δραστηριότητες, ε, ε, δραστηριότητες μάθησης κλπ. Μην ξεχνάμε ότι οι ηλικιωμένοι μπορούν να προσφέρουν πολλά και στο πλαίσιο της οικογένειας, εμπλεκόμενοι σε διάφορες δραστηριότητες, εθελοντισμού κλπ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της μεταρρύθμισης των των συστημάτων υγείας και των συνταξιοδοτικών συστημάτων θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι υποφελείται η κοινωνία από τις γνώσεις των ηλικιωμένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε Τάκουλα για αυτήν την ε, πολύ καλή παρουσίαση του θέματος γνωρίζεις ότι μπορούμε να κάνουμε πολλές ε, ωραίες δηλώσεις, ε, να παραθέτουμε τραγουδάκια, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ερχόμαστε και στην ουσία, στην πράξη. Ξέρετε λοιπόν πως από πλευρά αγωνιστικότητας ε, της ευρωπαϊκής οικονομίας μιλάμε όλο και περισσότερο για μια παράταση της ενεργού ζωής, του ενεργού βίου. Πέραν των 60-65 ετών Φυσικά μιλάμε για άτομα τα οποία είναι σε θέση να συνεχίσουν να εργάζονται και πρέπει να τα ενθαρρύνουν να το πράξουν. Τώρα, όταν ε, μιλάμε για ηλικιωμένους ή μάλλον για άτομα έμπειρα, αν θέλετε, χρειάζεται η εμπειρία αυτή να μπορέσει να χρησιμεύσει και να υποφεληθεί η κοινωνία της στη Φιλανδία. Ξέρετε ότι έχουμε ένα πρόβλημα σχετικά με την ε, διάλυση των οικογενειών. Ε, υπάρχουν άτομα τα οποία ζουν μόνα τους, ε, κοιτάξτε πολύ, από τα, τα πρόσωπα. Πολλά αυτά τα πρόσωπα ζουν σε οίκους ευγυρίας. Εδώ θα πρέπει να φροντίσουμε, να ενθαρρύνουμε αυτά τα άτομα να ασκήσουν κάποια δραστηριότητα στο πλαίσιο του εθελοντισμού. Εδώ έχουμε, έχουμε την μοναδική ευκαιρία για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε αυτούς τους ανθρώπους στην έκθεση. Ξέρω ότι θα υπάρξουν πολύ καλές ιδέες. Ευχαριστούμε πολύ. Thank, thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Δεν υπάρχει μετάφραση στα τσεχικά και τα σλοβακικά, οπότε θα μιλήσω αγγλικά. Θα προσπαθήσω. Ε, ξεκινώντας, ε, να ευχαριστήσω τον κύριο Κακούλα για την ε, έκθεσή του. ανέφερε πολλά σημαντικά στοιχεία τη σημασία του πολιτισμού, των αθλητικών δραστηριοτήτων, της ενεργού γύρανσης, της διαβίου μάθησης και των τεχνολογιών. Αυτά είναι τα σημεία που εγώ θεωρώ ως πιο σημαντικά. Κάποια σχόλια τώρα για αυτά, γιατί δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα υπόθηκαν. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν τα φυσικά κοινωνικά ωφέλη ε, που παίρνουμε από αυτούς τους ανθρώπους λόγω της εμπειρίας, της γνώσης τους, πράγματα που δεν ρυθμίζονται μέσω της ε, νομοθεσίας. Ε, κάποιες φορές θεωρούμε ότι τα άτομα αυτά πρέπει ουσιαστικά να δικαιολογήσουν ακόμα και την παρουσία τους κάτι που θεωρώ γελίο. Δεύτερον, ο κύριος Τακούλα ανέφερε ήδη στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την με τη χρηματοδότηση για τις ε, σχεδιασμένες ε, δραστηριότητες. Ε, ξέρουμε ότι η Κομισιόν στην πρότασή της δεν ζητά περαιτέρω χρηματοδότηση ε, κοιτά πώς θα τα κάνει όλα αυτά μέσα από διοικητικό επίπεδο και μέσα από δωρεές. Ε, συμφωνώ όμως με αυτό που είπε πριν ο κύριος Στακούλα ότι ειδικότερα σε εποχές ε, περικοπών ίσως να είναι δύσκολα τα πράγματα. Στην Τσεχία τουλάχιστον όταν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα ο πολιτισμός είναι το πρώτο που κόβεται. Και αυτός ε, πρέπει να είναι ο βασικός στόχος, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν ε, ουσιαστικά θεσπίζουμε αυτό το έτος ε, της ενεργού γύρανσης. Ε, Παρ' όλα αυτά χαίρομαι που μας φέρατε αυτό το σημαντικό θέμα εδώ ενώπιό μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κλάκια. Ευχαριστώ. Να συγχαρώ τον κύριο Τακούλα με τον τρόπο που χειρίστηκε το, το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για αυτούς να μείνουν ενεργοί στην ε, κοινωνία και να ε, συμμετέχουν είτε μέσω αποσχόλησης είτε μέσω εθελοντισμού, γιατί είναι μεγάλη συνεισφορά τους. Μίλαγα χθε με κάποιους φίλους, είναι οι φίλοι του Εθνικού ε, Μουσείου, είναι προστάτες ας πούμε του μουσείου και στην ουσία ε, βοηθούν και, την έβρεση, και για την, στην έβρεση κονδυλίων, ανταλλαγή μεταξύ σχολείων και τέτοια πράγματα. Είναι πολλά που μπορούν να γίνουν. Είναι μεγάλη ευκαιρία που έχουμε χρησιμοποιώντας τους ανθρώπους αυτούς και ακούγοντάς τους να κερδίσουμε εμπειρία. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, να πω ε, εγώ είμαι ήδη μεγάλη, δεν ξέρω αν θα δουλεύω εδώ τα επόμενα τρία χρόνια. Ε, η ενεργός ε, γύρανση παρόλα αυτά είναι δυνατή και απαραίτητη όπως βλέπετε. Στην τελευταία συζήτηση εγώ είχα ήδη πει ότι το, στο σημείο στην τροπολογία 2 θα ήθελα να να μιλήσουμε ξεκάθαρα για το senior service. Πολλοί από εμά μπορούμε να βοηθήσουμε με τις γνώσεις μας στην πολιτική ε, γυτνίασης, ε, ανάπτυξης κτλ. να συνεργαστούμε. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ξαφνικά από μάνατζερ βγαίνουν στη σύνταξη και από την εμπειρία μου βλέπω ότι στις χώρες ε, που δεν είναι τόσο ανεπτυγμένες, η λέξη senior service ε, και η δυνατότητα της χρήσης των ε, ηλικιωμένων στην πολιτική ανάπτυξη κτλ. είναι κάτι που πρέπει να δοθεί μέσα από αυτή την τροπολογία. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρετε ξεκάθαρο το πρόγραμμα αυτό στην τροπολογία. Να μιλάμε για διαβίου μάθηση μεν, αλλά να αναφέρεται και το γεγονός ότι το πρόγραμμα αυτό ουσιαστικά μέσα της διαβίου μάθησης μας φέρνει όλα αυτά που επιθυμούμε. Δηλαδή ε, μια επαφή με ιδέες κτλ. Νομίζω ότι αν γίνει αυτό θα είναι πλήρως ολοκληρωμένη η πρόταση και η, ε, και η έκθεση. Αν θες να πεις κάτι. Ε, μάλλον η Κομισιόν πρώτα. Ποιο από την Κομισιόν θέλει να μιλήσει, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από το 2008 υπάρχει μια γραμμή χρηματοδότησης ε, για, τις ε, εθελοντικές, ε, για τα εθελοντικά σχέδια για την γύρανση για τους ηλικιωμένους. Είναι 1,5 δις ευρώ Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες που ουσιαστικά προσφέρονται μέσα από αυτό το κονδύλι και είναι πολλά τα project. Στην εξάντια αξιολόγηση αναφέρονται συγκεκριμένα στοιχεία από την Κομισιόν και υπάρχει και μια σειρά δραστηριοτήτων ε, επαιτειακού χαρακτήρα, ε, ας πούμε κάποιες ε, τελετές έναρξης και λήξης. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα χρήματα. Μπορούμε να δώσουμε λοιπόν τους πόρους για να χρηματοδοτηθούν σημαντικές δραστηριότητες. Ε, όντως αναγνωρίζω το σημείο που ανέφερε η κυρία Κάτζαν για, τους εθνικούς, ε, για τις εθνικές περικοπές στους προϋπολογισμούς. Ε, όντως, ε, όταν υπάρχει αυτή η υποχρέωση συγχρηματοδότησης, ίσως οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται να μην είναι τόσο πολύ, πολλές. Έγινε όμως μια συνάντηση με τους ε, εθνικούς συντονιστές στις Βρυξέλλες και πριν ε, εγκριθεί επισήμως αυτό το ευρωπαϊκό έτος, γιατί θεωρούσαμε ότι όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα. Τώρα έχουμε και συναντήσεις με τους εθνικούς ε, φορείς για να μπορέσουμε να οργανώσουμε όσο περισσότερες δραστηριότητες γίνεται. Ευχαριστώ. Χάνω τώρα. Έχεις το λόγο. Arvoisa puheenjohtaja, kun lopetin Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προλίγου αναφέρθηκα σε ένα φιλανδικό τραγούδι και άκουσα τα λόγια σας πρόεδρε και μου έρθει στο μυαλό ένα άλλο φιλανδικό τραγούδι που φέρει τον τίτλο Doris. Doris, Doris, ε, πραγματικά με συναρπάζεις. Και λοιπά και λοιπά. Με στόση πάντως ε, είμαι πρόθυμος ε, να δεχτώ αυτή την προσθήκη την οποία αναφέρατε στο, στο κείμενό μου. Να πω εξάλλου ότι όλα όσα ακούστηκαν ε, ε, ε, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Πραγματικά οριμάζουμε με τρόπο ενεργό θα έλεγα. τώρα αυτό το οποίο προέχει είναι να καταλήξουμε σε μια γνωμοδότηση ως το δυνατόν καλύτερη. Τώρα, σε ό,τι φορά τα οικονομικά, τα δημοσιονομικά ζητήματα, νομίζω πως ο Μάρτιν Κάσλερ ε, ασχολείται με αυτά. Εμείς θα πρέπει να ασχοληθούμε με την πολιτική πτυχή του ζητήματος. Δηλαδή αυτό που εμπίπτει από όλες τις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου πρέπει να καταθέσετε τις τροπολογίες σας. Ε, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, 9 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ Χανό και αγαπητοί συνάδελφοι. Ερχόμαστε τώρα στο σημείο 10, νεολαία σε κίνηση, μια πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων των νέων με στόχο την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς επιπλέον χρήματα. Κύριε Τσβέρ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Όλοι. Όλοι είναι νέοι. Ε, θέλω να πω ότι αυτό το οποίο τώρα σα λέω είναι συνέχεια τη γνωμοδότησης που ακούσαμε τον κύριο Τάκουλα. Όλοι είμαστε νέοι και η διαφορά είναι ότι ορισμένοι είναι νεότεροι από του άλλου ή κάποιοι λιγότερο από του άλλου. Και για να προσθέσουμε κάτι σε αυτό το οποίο ελέγχθησαν, αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι οποιοδήποτε ηλικιωμένο να έχει την ευκαιρία να μπορεί να συνεχίσει να παρακολουθεί ό,τι τον ε, ενδιαφέρει. Ε, αλλά αυτό είναι σημαντικό και για την κοινωνία γενικότερα, να μπορούν επομένω οι ηλικιωμένοι να μην περιθωριοποιούνται στην κοινωνία. Και γι' αυτό και σας λέω ότι θα πρέπει να έχουμε ε, ενεργούς πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας. Τώρα για αυτή την ε, πρωτοβουλία να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή σας, την Επιτροπή μας μάλλον, γιατί έτσι έχω την ευκαιρία να μιλήσω πάνω σε αυτό το σημαντικό θέμα. Βεβαίω και ε, το, υπάρχει θέμα χρηματικό, αλλά θα το συζητήσουμε καλύτερα. Και όσον αφορά κάποιο σκεπτικισμό θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να αποφευθεί ε, η ιδέα αυτή να ξαναμείνει ένα κενό γράμμα. Εγώ έχω μελετήσει τους ε, στόχους και συνειδητοποίησα ότι αυτή η πιλωτική πρωτοπόρο πρωτοβουλία την επόμενη δεκαετία θα είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτό κυρίως όσον αφορά την ε, στρατηγική για το 2020 και τους στόχους της. Πρώτα πρώτα να πούμε δύο λόγια όσον αφορά την ανταλλαγή των απόψεων για την πρωτοβουλία η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη. Πρώτα πρώτα παιδεία εκπαίδευση και κατά δεύτερο λόγο έχουμε το θέμα της ε, απασχόλησης των ε, νέων. Βεβαίως, ε, απασχόληση είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει την Επιτροπή, την Αρμόδια. Αλλά είναι κάτι που συνδέεται άρρηκτα και με τη δική μας αρμοδιότητα. Για να δούμε τώρα. Ο βασικός στόχος της υπόθεσης αυτής είναι το να μπορέσουμε να προσδώσουμε τους ε, νέους την ε, γνώση, τη γνώση που θα τους ε, επιτρέψει να μπουν στην αγορά εργασίας και να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τις μεταρρυθμίσεις της αγοράς απασχόλησης. Δεν έχουμε κάποιο κονδύλιο το οποίο πρικοδοτεί αυτή την ιδέα. Όμω υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Δύο λόγοι. Πρώτα πρώτα η πρωτοβουλία έχει σχέση με το πρόγραμμα που τώρα τρέχει και που την χάνει πρικοδότησης. Οπότε κομισιόν και οι άλλες υπηρεσίες επιμελούνται της συνέχισης του πρόγραμματος που τώρα τρέχει. Θέλουμε να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτής της πρωτοβουλίας και της πρωτοβουλίας για την ε, ισόβια κατάρτιση, μάθηση. Μήπως εδώ έχουμε κάποιο επικάλυψη, έστω και μερική, που είναι αρνητική. Γιατί η ισόβια κατάρτιση έχει προοικοδότηση, έχει προσωπικό που ασχολείται με αυτή την ιδέα, ενώ η πρωτοβουλία την οποία τώρα συζητούμε για τους νέους είναι μια πνοή δροσερού αέρα, μπορούσε να πει κανείς. Είναι κάτι το φρέσκο, κάτι το καινούριο, το οποίο πρόκειται να είναι αέρα στα πανιά ε, αυτών που ωφελούνται από την πρωτοβουλία. δεν ξέρουμε κατά πόσον ε, αυτή η πνοή θα έχει την απαραίτητη ισχύ. Άρα θα πρέπει να ε, ψάξουμε περισσότερο το θέμα. Είναι τμήμα της στρατηγικής για το 2020 και είναι πολύ σημαντική. Η στρατηγική αυτή βέβαια έχει στόχο το να μπορέσουμε να έχουμε μια ευφυή και βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλουμε την απασχολησιμότητα του ενεργού πληθυσμού. Να πάμε στο 69, στο 75% από 1,9 να πάει 3% του ΕΠ, ε, το χρήμα το οποίο αφιερώνεται στην έρευνα και επίσης από το 31% από 40% το ποσοστό των νέων που έχουν προστιμιακά διπλώματα. Να σταματήσει επίσης ε, ή τέλος πάντων να πέσει από το 10% μάλλον να πάει 10% από 15% το ποσοστό αυτών οι οποίοι εγκαταλείπουν την παιδεία. Από 80 εκατομμύρια πάμε σε 60% ε, αυτούς που μαστίζονται από τη φτώχεια και να καλύψουμε, είπαμε κυρίως τους νέους, να ε, κινηθούμε στα πλαίσια αυτής της σημαντοπιστωτικής κρίσης και να δούμε το ότι από 20% ανέβηκε σε 21% η ενεργεία για τους νέους. Έχουμε 5 εκατομμύρια νέους οι οποίοι δεν έχουν δουλειά. Δηλαδή, δύο φορές τον πληθυσμό της χώρας μου, της Σλοβενίας. Τόσοι είναι οι άνεργοι νέοι. Και λέει η επισημότητα ότι ακόμα και σε περίοδο ε, κρίσης και αρνητικού ρυθμού ανάπτυξης Ακόμα και τώρα υπάρχουν θέσει εργασία που δεν έχουν καταληφθεί. Και από την άλλη όμω έχουμε νέου που δεν μπορούν να βρουν δουλειά γιατί δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Επομένω, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τι ιδέε μα όσον αφορά τα συστήματα εκπαίδευση και κατάρτιση. Με λίγα λόγια, πάνω από αυτά τα συστήματα είναι ανεπαρκή για τι ανάγκε τη Ευρώπη. Και για αυτό και αναλαμβάνονται αυτές οι πρωτοβουλίες, ούτω ώστε αυτά τα συστήματα κατάρτισης και εκπαίδευσης να προσαρμοστούν στις ανάγκες αγοράς εργασίας. Φυσικά θα πρέπει να φροντίσουμε και την κινητικότητα των νέων, να προσαρμοστούν και αυτοί στις ανάγκες της κοινωνίας. Οπότε, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία αφορά και τη μάθηση αλλά και την απασχόληση. Δεν περιορίζεται στην ανταλλαγή καθηγητών, φοιτητών, μαθητών κλπ. Αλλά προβλέπει έναν μηχανισμό για να βελτιωθεί η παιδεία και η εκπαίδευση των νέων και έτσι να μπορούν οι νέοι, εκτό από την παιδεία, να μπορέσουν και πλευρά πολιτιστική να ωφεληθούν. Δηλαδή να, μπορούν, να μπορεί τελικά πραγματικότητα να πλησιάσει στα εκδοτικά συστήματα και αντιστρόφω. Έχουμε εδώ πολλέ επιμέρους ε, ιδέες για αυτή την πρωτοβουλία. Ε, πάντοτε βέβαια έχονται βελτίωση αυτέ οι προτάσει. επαγγελματική κατάρτιση, ήδη έχουμε ε, κάποιες πρωτοβουλίες που την καλύπτουν, έχουμε συστήματα αξιολόγησης για τα πανεπιστήμια, όλα αυτά ε, αποτελούν αντικείμενο κοινωτικών προγραμμάτων εδώ και μια δεκαετία και παραπάνω και ε, τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα μάλλον πετυχημένα είναι. Έχουμε και την διαδικασία της Μπολόνια ε, που βεβαίως είχε κάποιες διασυπτώσεις, αλλά η Μπολόνια, η πρωτοβουλία αυτή σημαίνει περισσότερα ε, πράγματα. Ε, δηλαδή θέλω να πω ότι θα πρέπει πέρα από τα πανεπιστήμια η διακρισία της Μπολόνια να ωφελήσει και τα χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης. Θέλουμε το 2020 ή μέχρι το 2020 το 50% των επαγγελμάτων να να επανδρώνονται κατά κάποιο τρόπο με αποφύτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και αποφύτους πανεπιστημίων. Άλλαξαν τα πράγματα περισσότερο από όσο περιμέναμε όταν φτιάξαμε την διαδικασία της Μπολόνια. Άρα πρέπει να καλύψουμε τώρα όχι μόνο το πανεπιστήμιο αλλά όλα τα, τα, επίπεδα ε, στην κλίμακα της παιδείας, στην πυραμίδα της παιδείας μέτρα χρειάζονται, δράσεις χρειάζονται ε, και εγώ σας αναφέρω μερικά γιατί χρειάζονται και άλλα πράγματα όπως ας πούμε κάποιο website το οποίο να αφορά μόνο αυτή την πρωτοβουλία ε, για την απασχόληση, άλλο website όσον αφορά το παρατηρητήριο για την κατάρτιση και όσον αφορά την κινητικότητα θα έχουμε ένα πίνακα αξιολόγηση και μια βάση δεδομένων. Και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα κληθεί να καλύψει με πιστώσεις και με δάνεια την κινητικότητα των νέων. Πάντως, κινητικότητα δεν σημαίνει μόνο γνώση ξενογλωσσών. Σημαίνει και οικονομική δυνατότητα οικονομική υποστήριξη. Γιατί πολλές φορές οι νέοι που προέρχονται από φτωχότερε περιοχές τη Οικονομικής Ένωση έχουν λιγότερα χρήματα, δηλαδή είναι λιγότερο κινητικοί. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα βοηθήσει πάρα πολύ σημαντικά με τα χρήματα που θα δώσει την υπόθεση της κινητικότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει το δικό της σύστημα αξιολόγηση πανεπιστημίων στο μέλλον. Είναι κάτι αυτό το οποίο χρειάζεται. Λείπει εδώ και πολύ καιρό. Γιατί τα δεδομένα που έχουμε δώσει διάθεσή μας είναι πάρα πολύ φτώχα. Χρειάζεται επομένω μια αξιολόγηση, μια βαθμολόγηση των πανεπιστημίων που να είναι αξιόλογη, πάρα πολύ σημαντικό και τα πανεπιστήμια δεν είναι δυνατόν να αξιολογούνται μόνο με λίγα και κάπως αυθαίρετα κριτήρια. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσον χρειάζεται να αναπτύξουμε κάποια κάρτα, ειδική κάρτα. Αυτή η κάρτα που θα αφορά το τρέχον πρόγραμμα θα συμπληρώσει τις υπάρχουσες κάρτες και ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή όλες οι κάρτες να γίνουν μία. Είπαμε ότι δεν έχουμε κονδύλια για την πρωτοβουλία αυτή. Όμως, η επιτυχία εξαρτάται από την προοικοδότηση. Μέχρι το 2013 ή μέχρι το 2030 δεν θα μπορέσουμε να έχουμε την ανάλογη κάλυψη, αλλά ίσως μετά. Πάντως, εδώ έχουμε κάποια πάρα πολύ σημαντικά προγράμματα, Μαρία Κιουρί, Έρασμος και άλλα, και αυτά τα προγράμματα θα συνεχίσουν να έχουν την προοικοδότηση στο μέλλον και έτσι θα έχουμε καλύτερη κινητικότητα. Συχνά αναφέρεται ότι το 2020 όλοι οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν το εξωτερικό. Ίσως αυτό είναι λίγο υπερβολικό, αλλά μια που υπάρχει τώρα η τάση αύξησης κάποιων κονδυλίων, Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω αν είναι εύκολο να καλυφθεί αυτός ο στόχος και η χρηματοδότηση της ανταλλαγής μαθητών και σπουδαστών θα πρέπει να αυξηθεί αν θέλουμε να είναι πιο ευρωπαϊκά τα συστήματα παιδείας, κατάρτισης, εκπαίδευσης. Δεν μακρηγόρησα ελπίζω πρόεδρε, αλλά σας τονίζω ότι πρόκειται για κάποια πάρα πολύ θετική πρωτοβουλία. Μία φρέσκια πνοή όσον αφορά τα συστήματα παιδεία στην Ευρώπη. Mange tak, formand. Uh, undskyld, jeg sådan, uh, trænger mig på som en anden taler her, men jeg skal til møde her kl. 10, så jeg håber, at det er i orden. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μια συνεδρίαση στις 10 και θα χρειαστεί να, να χωρίσω. Ε, πολύ δύσκολο κανείς να διαφωνήσει με την υποεξέταση πρόταση. Είναι μια πρόκληση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Κατά τα υπόλοιπα συμφωνώ με πολλά από τα όσα ακούστηκαν. Θα ήθελα να επικεντρωθώ επί και μόνου θέματος σε αυτή την πρώτη αλλαγή απόψεων, ε, τη συνεργασία ανάμεσα στα πανεπιστήμια και τον ε, επιχειρηματικό κόσμο. Ε, Είμαι πολύ ικανοποιημένο από τι πρωτοβουλίε που προτείνει ο εισηγητή. Η ποιότητα τη συνεργασία ανάμεσα στα πανεπιστήμια και τον επιχειρηματικό κόσμο ε, θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, χρειάζεται να υπάρξει περαιτέρω εξυγχρονισμό αυτή τη σχέση και να δημιουργηθούν πραγματικέ εταιρικέ σχέσει. Το ζήτημα τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων που θα τεθεί ω τον ούπο δεν ε, αποτελεί μυστικό. Όλο και περισσότερε ιδιωτικέ ε, χρηματοδοτήσει γίνονται προς τα πανεπιστήμια, διότι το δημόσιο έχει αρχίσει τι περικοπές. Θα χρειάζεται λοιπόν σε αυτό να υπάρξει καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στα πανεπιστήμια και τον κόσμο τη οικονομίας. Υπάρχουν ε, φυσικά και μία σειρά από πολιτιστικούς φραγμούς ανάμεσα στα πανεπιστήμια και τον κόσμο της οικονομίας χρειάζεται να μιλούν όλη την αυτή γλώσσα. Δεν ε, πρέπει λοιπόν ε, να το παραμελήσουμε αυτό το ζήτημα σε ό,τι φορά τώρα τα πανεπιστήμια. Ξέρουμε ότι έγινε σημαντική πρόοδος στο πλαίσιο της αξιολόγησης των πανεπιστημίων πρέπει να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση από τα πανεπιστήμια. Θεωρώ πως ε, χρειάζεται να γκρεμίσουμε τα, όλους τα εμπόδια φραγμούς που υπάρχουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια πρόταση προκειμένου να προαχθεί η κατάρτιση των νέων και πέδες των νέων πρέπει να ρίξουμε τους φραγμούς που εμποδίζουν την κινητικότητα των νέων βλέπουμε ότι οι πίνακες παρακολούθησης που έχουν δημιουργηθεί αποτελούν ένα πολύ ικανοποιητικό μέσο για την βελτίωση των, της καταστάσεως Τώρα κάτι ακόμα που μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές. Δεν ε, θα πρέπει να ξεχνάμε πως το 5% των ε, δανών ε, νέων εκπαιδεύονται στο τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό εντάξει δεν είναι στα πλαίσια της Επιτροπής μας αυτό καθε αυτό, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε πώς ε, θα μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και αυτά τα άτομα στην έκθεσή μας. Αυτά είχα, έχω να πω προς το παρόν και να πω ότι με ικανοποιεί η έκθεση αυτή του εισηγητή. Ευχαριστώ. Να σας πω ότι η Επιτροπή Απασχόλησης ε, έχει ε, ίδια, συμμετοχή με εμάς. Εμείς κάνουμε τη δική, τους, τη δική μας συμβολή και μετά οι δύο εισηγητές θα συζητήσουν, έχουν συζητήσει μάλλον και ήδη, αλλά θα συζητούν εντατικά και κατά τη διάρκεια των εργασιών και των δύο ε, επιτροπών, γιατί και η Επιτροπή Απασχόλησης είχε ενδιαφέρον λόγω της επαγγελματικής κατάρτισης που εμπλέκεται στην έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ε, ζητώ συγγνώμη που άργησα και άκουσα μόνο το τελευταίο κομμάτι της ε, παρουσίασης. Παρ' όλα αυτά, έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχάς, σε επίπεδο κινητικότητας υπάρχουν πολλά προβλήματα που υπάρχουν και ήδη έχουν αναφερθεί, όμως υπάρχουν και κάποια άλλα που θέλω να αναφέρω και έχουν να κάνουν με τη ε, διαδικασία της Μπολόνια. Ακούω συνεχώς από φοιτητέ που θέλουν να πάνε στο εξωτερικό ότι λόγω των επιπτώσεων της διαδικασίας της Μπολόνια έχει γίνει όλο και πιο δύσκολο να το κάνουν αυτό. Είναι δύσκολο ε, να αναγνωρίσουν στο δικό τους πανεπιστήμιο ε, τα πιστοποιητικά που παίρνουν σε ένα άλλο πανεπιστήμιο και έτσι ε, χάνουν το εξάμεινό τους. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, Ε, μέσα από τη διαδικασία της Μπολόνια ε, κάνει την φίτηση γενικότερα πολύ δύσκολη ε, και την εμποδίζει πολλές φορές. Έτσι λοιπόν τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιγόντως να ξανασκεφτούν τη διαδικασία της Μπολόνια με τέτοιο τρόπο ώστε να τη διαμορφώσουν να τη διαμορφώσουν μάλλον με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζει την κινητικότητα. Πραγματικά δεν ξέρω αν πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήταν λογικό ε, αν, ε, για παράδειγμα, είχαμε ένα website όπου ε, οι νέοι θα μπορούσαν γρήγορα να δουν τι μπορούν να που μπορούν να φοιτήσουν σε ποιο πανεπιστήμιο, ποια μαθήματα θα βρουν εκεί και να παρατίθενται όλα τα πανεπιστήμια με τη σειρά. Θεωρώ ότι αυτό ε, θα ήταν χρήσιμο όπως επίσης ε, να αναφέρεται ποιο είναι το καλύτερο ή το χειρότερο πανεπιστήμιο στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν ε, σε κάθε τομέα, σε κάθε ειδικότητα θα μπορεί κανείς να βρίσκει ποιο είναι το καλό και το κακό πανεπιστήμιο και πραγματικά νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να ξανασκεφτούμε γιατί συνεχώς ακούω παράπονα και ε, μια τέτοια μορφή σκέψης και επιλογής θα μπορούσε να βοηθήσει τους νέους που συνεχώς συζητούν αυτό το θέμα και νομίζω ότι στην Επιτροπή μας είμαστε σύμφωνοι ότι το Youth on the Move είναι ένα πρόγραμμα που θα πρέπει να έχει επιτυχία σε επίπεδο ε, εκπαίδευσης ε, και κατάρτισης θα μπορούσε λοιπόν να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Διότι ακούμε για το Youth on the Move, έχουμε δημιουργήσει ε, κάποια προϊόντα αναγνωρίσιμα στην Ευρώπη και είναι καλό κανείς να μπορεί να τα αναγνωρίζει και να συνδέεται με αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βάρκο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητή Επιτροπή. Η φιλανδογκρική παράδοση επιτάσσει να τραγουδάμε λαϊκά τραγούδια, παραδοσιακά τραγούδια. Όμως εγώ από την, από την πλευρά μου θα ήθελα μάλλον να αναφερθώ στο γεγονός ότι το θέμα για το οποίο συζητάμε σήμερα είναι ένα θέμα που θα αντιμετωπίσουμε και θα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα 25 χρόνια. Μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό όνειρο, για ένα σλόγγαν ε, ε διαφορετικότητας και τα λοιπά που χρησιμοποιείται συνεχώς ε, εδώ στο ε, κοινοβούλιο. Το σχετικό τραγούδι που μου έρχεται στο μυαλό είναι το Papa Don't Preach της Μαντόνα. Γιατί εμείς δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα των νέων αν δεν τους ε, κάνουμε να συμμετάσχουν και αυτοί σε αυτή τη διαδικασία. Συνήθως ε, οι νέοι αμφισβητούν τις αλήθειες που τους περνά η μεγαλύτερη γενιά ως δεδομένες. και είναι πιο στενά συνδεδεμένη με το σημείο της ημερήσια διάταξη νούμερο 10 από ότι εμεί. οι περισσότεροι από εμά νομίζω. Αντί λοιπόν να απελευθερώσουμε απλώς το δυναμικό των νέων, ε, απελευθέρωση δηλαδή, αντί για τον όρο απελευθέρωση, καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη λέξη, μια άλλη ορολογία. Ίσως να μιλάμε καλύτερα για υποστήριξη βοήθεια, αρρωγή, ε, όχι απελευθέρωση του δυναμικού. Έτσι λοιπόν θα ήθελα μάλλον να κάνω μια τροπολογία με αυτό το στόχο. Όσοι μίλησαν, μίλησαν για, πριν από μένα, μίλησαν για τη σημασία του θέματος, ε, για το θέμα της κινητικότητας, που πραγματικά και εγώ υποστηρίζω, όμως και ένα άλλο θέμα το οποίο ε, συχνά συζητείται είναι το πρόγραμμα Εράσμους που θα έπρεπε και αυτό να βρίσκεται σε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης, σε αυτό το θέμα μας. Ε, δεν αναφέρεται, τουλάχιστον στη διάσταση που ήθελα εγώ, να υπάρχει ένα εράσμος για τον αθλητισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κ. Μάρκος Κορέα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο Σουάμπ για την ε, πρώτη έκθεση που αφορά στην ε, πρωτοβουλία αυτή για την διαλύση κίνηση. Δεν ξέρω αν ε, πράγματι κάναμε χάρη που το αναθέσαμε αυτή την έκθεση, διότι είναι μια έκθεση ιδιαίτερα σημαντική μεν, αλλά και ιδιαίτερα περίπλοκη και προβληματική. Διότι αφενός γνωρίζουμε δεν υπάρχει συγκεκριμένη γραμμή του προπολογισμού και άρα όλα όσα μπορούμε εμείς να προβλέψουμε χρειάζεται να δούμε πώς ε, θα μπορέσουν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέγεται ότι πρόκειται για μια ευληματική πρωτοβουλία και φυσικά κάνει κάποιες προτάσεις, αναφέρει κάποιες σκέψεις, προβληματισμούς κλπ. Ε, στο πλαίσιο των οποίων ε, φαντάζομαι πως συμπεριλαμβάνονται τα πολιετή προγράμματα για την νεολαία, για τα οποία φυσικά έχουν ε, χρηματοδότηση και άρα δεν θα πρέπει, θα πρέπει να προσέξουμε να μην υπάρξει επικάλυψη, να μην γίνουν παρανοήσει ε, και να μην υπάρξουν περαιτέρω περικοπές στον προπολογισμό επειδή υπάρχει μια νέα πρωτοβουλία και να αφαιρεθούν κονδύλια από, άλλες, ε, από άλλα προγράμματα. Και χθε στο πλαίσιο των συντονιστών εξέφρασα κάποιε ανησυχίε, διότι στην ε, ανακοίνωση τη Κομισιόν επί του προγράμματο εργασία για το προσεχέ έτο που αφορά στα πολιετή προγράμματα για τη νεολαία θα πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν ποιο θα είναι το εύρος αυτής της ε, Πρωτοβουλία νεολαία σε κίνηση. Ελπίζω ακόμα και σήμερα η Κομισιόν να μας δώσει κάποιες περαιτέρω διευκρινήσει. Τώρα σε ό,τι αφορά το κείμενο αυτό καθεαυτό θα έχουμε και άλλε ευκαιρίες για ανταλλαγή απόψεων. Σημασία έχει να συμπεριληφθεί όλο το ζήτημα της απασχόλησης, όλος ο σχετικός προβληματισμός, διότι αυτή την περίοδο κρίσης χρειάζεται να υπάρξουν ιδιαίτερα στηρίγματα στους νέους διότι φορά την εξέβριση εργασίας. Προς το παρόν μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα το ζήτημα, αλλά ο, οι νέοι δεν ε, έχουν επωφεληθεί ιδιαίτερα. Πρέπει να ε, εξεταστεί περαιτέρω το ζήτημα. Ο συνάδελφος ε, Σουέρ ε, σίγουρα θα το θα το θίξει το ζήτημα. Αυτός είναι πολύ, πολύ χρήσιμη αυτή η πρώτη αλλαγή απόψε. Ευχαριστώ Μάρκο. Τελευταία μιλήτρια κυρία Μακλάρκεν. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να λάβουμε υπόψη μας την οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να επικεντρωθούμε στις ε, προτεραιότητες. Το 40% ο ε, στόχος για το πανεπιστήμιο δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει. Ε, προσπαθήσαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, είμαι όχι τόσο μεγάλη επιτυχία. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε, <clears throat> να επιμείνουμε στην ευέλικτη μάθηση, να δούμε τι γίνεται με τους νέους που δεν θα πάνε στο πανεπιστήμιο, να υπάρχουν ε, στην αγορά ευέλικτα ε, συμβόλαια και θέσεις εργασίας, ε, γιατί υπάρχουν οι δεξιότητες που θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω κι εγώ κάτι αυτά που είπε η κυρία Μακλάρκινγκ, συμφωνώ. Χθε είχαμε μιλήσει για την επαγγελματική κατάρτιση και μάθηση και θεωρήσαμε ότι αυτό το θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης θα πρέπει να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν είναι 40% όλοι αυτοί που θέλουν να τελειώσουν και μπορούν να τελειώσουν το πανεπιστήμιο. Όχι μόνο λοιπόν 40% πτυχίο πανεπιστημίου, αλλά πτυχίο πανεπιστημίου ή κάτι παρόμοιο, μια επαγγελματική κατάρτιση. Κάτι ισότιμο, κάτι ισότιμο μάλλον. Η επαγγελματική κατάρτιση είναι πολύ σημαντική. Πρέπει και αυτός ο τομέας να ενισχυθεί. Αυτοί που παίρνουν το απολυτήριο του ε, σχολείου θα πρέπει μετά να μπορούν να ε, συμμετέχουν σε μια τέτοια επαγγελματική κατάρτιση, διότι χρειαζόμαστε και τέτοιους ανθρώπους, πολύ περισσότερο από ό,τι ε, μπορείτε να φανταστείτε. Έτσι λοιπόν, 40% άτομα με ανώτατη εκπαίδευση ή κάτι ισότιμο. Επίσης, για το ranking. Ε, θα απορούσα αν έκανε η Κομισιόν ένα τέτοιο ranking. Ε, πραγματικά δεν θα γίνει τίποτα. Μπορεί να το προσπαθήσει, αλλά αν θυμάστε στο παρελθόν, ε, προσπαθήσαμε πριν από την κύριε Βασιλείου να το κάνουμε αυτό και τελικά δεν πέτυχε. Πρέπει πραγματικά να σκεφτούμε ότι θα ήταν λάθος. Μια πύλη ίσως θα ήταν ε, μια λύση, αλλά θα ήταν λάθος να πάμε πιο συγκεκριμένα σε ranking. Πώς θα γίνει από τη Ρωμανία μέχρι την Πορτογαλία είναι τρελό, δεν ξέρω, δεν μπορούμε να το δούμε τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι σωστή η άποψη που έχουμε γι' αυτό. Σε μας δεν θα γίνει, σίγουρα. Τώρα για την νεολαία. Κι εγώ δεν ανήκω στην νεολαία πλέον. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν με ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Έχω παιδιά, έχω εγγόνια και ξέρω ποιε είναι οι ελλείψεις. Είναι δική μας λοιπόν η ευθύνη να έχουμε μια καλή ε, πολιτική για τους νέους, τους οποίους να ανήκουμε. Το Φόρουμ των Νέων είναι κάτι ε, που είναι το αντίστοιχο των δομών της Κομισιόν. Γίνονται προτάσεις στην Κομισιόν, ακούγεται αυτό το Φόρουμ και νομίζω ότι είναι καλό να δώσουμε μια φωνή στους νέους σε αυτό το θέμα. Τώρα για το Youth on the Move. Και αυτό είναι μια αναβαρχίδα με μια έκθεση πολύ σημαντική. Δεν ξέρω όμως πώς θα λειτουργήσει. Γιατί έχει ξεραθεί η θάλασσα και δεν μπορεί να προχωρήσει το πλοίο. Και δεν ξέρουμε καν τι υπάρχει μέσα σε αυτό. Δεν είναι καν πρόγραμμα. Δεν πρέπει να είναι πρόγραμμα, είπαμε γιατί έχουμε προγράμματα όπως το Εράσμους, το Κορμένους, όλα αυτά είναι προγράμματα που είναι γνωστά, τα γνωρίζει ο κόσμος και τρέχουν. Το Youth on the Move είναι απλώ μια ιδέα που θα υποστηρίζει ακόμα περαιτέρω αυτά τα προγράμματα και θα τους δίνει μεγαλύτερη σημασία. Έτσι λοιπόν, ε, σας προειδοποιώ στην Κομισιόν να μην κοιτάτε μας από τα μάτια των Βρυξελών, ε, μόνο και να μην το κάνετε σαν ένα μεγάλο πρόγραμμα. Εγώ δεν θα συμφωνήσω. Δεν βλέπουμε καν τα πολιτή προγράμματα εκεί, στην Κομισιόν. Έχουν εξαφανιστεί. Ε, Γι' αυτό το λόγο λοιπόν όσοι είστε εδώ από την Κομισιόν να σας πω να μεταφέρετε στους ανωτέρους σας ότι η Επιτροπή μας δεν θέλει αυτό το πρόγραμμα ε, το Youth on the Move να κάνει όλα τα υπόλοιπα προγράμματα που τρέχουν να καταρρεύσουν. Θα ζητήσω λοιπόν από την Κομισιόν να προσπαθήσει αναξάρτητα με το πόσα χρήματα θα πάρουμε, πόσα λίγα χρήματα ή πόσα λίγα ε, γνωρίζουμε, να μην ε, συζητούμε προς αυτή την κατεύθυνση. γιατί θα πάμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο στο Συμβούλιο. Εμείς θέλουμε δομημένα προγράμματα, δομημένο εράσμους, κορμένους κτλ. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Για μένα λοιπόν είναι ύποπτο αυτό το θέμα. Κανέναν δεν εμπιστεύομαι, ούτε καν την Κομισιόν. Γιατί βλέπω ότι εκ των προτέρων κάνει κάτι αποτρόπαιο για μένα. Κάτι που δεν μπορώ καν να φανταστώ. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι εργαζόμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Θέλει να μιλήσει παρ' όλα αυτά. Ναι. Όχι. Ναι. Who wants, who wants to... Ποιος θέλει να μιλήσει. Θα τολμήσετε. Ορίστε. Okay, thank you very much, um, President. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ επίσης ε, και τα αξιότιμα μέλη για το όσα ανέφεραν σχετικά με το ζήτημα. Θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για μια ευλυμπατική πρωτοβουλία για τη στρατηγική του 2020 και είναι πολύ σημαντικό να προωθήσουμε την εκπαίδευση και την κατάρθεση για θέματα απασχόλησης των νέων όπως αναφέρει και η Κομισιόν και προσέθεσε αυτή ως μία από τις 7 ε, εμβληματικές πρωτοβουλίες. Μιλάμε εδώ για μία στρατηγική. Πρόκειται για μία ατζέντα που περιέχει μία σειρά πρωτοβουλειών. Ορισμένες από αυτές έχουν ήδη παρουσιαστεί, άλλες ε, θα παρουσιαστούν τα προσεχή έτη. Πρόκειται για δράσεις ε, κλειδί Προτείνουμε όμω επίση να ενισχύσουμε κάποιες ήδη υφιστάμενε δραστηριότητε. Θέλουμε να προάγουμε επίση και τι ε, πρωτοβουλίε αυτές. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πω πρόκειται για μια στρατηγική, μια ατζέντα πολιτικών και στρατηγικών. Εδώ δεν ε, αναφερόμαστε σε όλες τις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο θέμα της απασχόλησης. Αφορά αυτή η πρωτοβουλία μόνο τους νέους. Και ένα από τα σημεία κλειδί αυτής της ε, ατζέντα είναι ότι συνδυάζεται με το τι θα συμβεί μετά από το πέρας ε, των σπουδών. Συνδέεται λοιπόν άμεσα με τον χώρο της ε, εργασίας. Λοιπόν, όπως είπατε, όχι μόνο σε αυτή την πρωτοβουλία, αλλά και στη στρατηγική της ε, Ευρώπης 2020 υπάρχουν πολλές δεσμεύσεις από πλευρά της και του Συμβουλίου, αλλά και του Κοινοβουλίου, αναφορικά με την σημασία της ε, κοινοτικότητας στην εκμάθηση Υπάρχει λοιπόν μεγάλη προσπάθεια σε αυτό το θέμα όπως και στη μεταρρύθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Να πω επίσης ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές στηρίζονται από πολλές δράσεις. Είπε η κυρία Πακ το θέμα των προγραμμάτων εκπαίδευσης κατάρτισης. Όταν μιλάμε για κινητικότητα της μάθησης, ε, έχουμε το πρόγραμμα της νεολαίας εκκίνηση και υπάρχει και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες λοιπόν χρηματοδότησης από διάφορα ταμεία του των λεχθέντων λοιπόν θα ήθελα να αναφερθώ ότι η νεολαία σε δεν είναι το παν. Αυτή η πρωτοβουλία συμπληρώνει τις ίδιες υπάρχουσες. Υπάρχουν, υπάρχει το ευρύ στρατηγικό πλαίσιο που ενέκριναν οι Υπουργοί το 2009 σχετικά με την συνεργασία και την εκπαίδευση και κατάρτιση και η νεολαία σε κίνηση δεν θα αλλάξει φυσικά όλα αυτά τα προϋπάρχοντα. Κτίζουμε λοιπόν πάνω στα ήδη υπάρχοντα και εστιάζουμε στην ε, πρωτοβουλία αυτή σε θέματα που αφορούν ε, τους νέους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Τώρα, επανέρχομαι στο ζήτημα της χρηματοδότησης. Ε, όπως γνωρίζετε, είναι πολύ κρίσιμη περίοδος για το ότι θα έχουμε στα επόμενα προγράμματα. Έχουμε διαμόσια διαβούλευση, η οποία ξεκίνησε την ίδια μέρα που ξεκίνησε και η νεαλία σε δράση έγινε μια δημόσια διαβούλευση για το σύνολο των προγραμμάτων για μετά το 2014. Έχουμε, είχαμε διαβούλευση για την νεολαία σε κίνηση, για την διαβίου για το έρασμος κλπ. Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε πριν από δύο ημέρες με ένα πολύ ψηλό αριθμό απαντήσεων, πάνω από χίλιες απαντήσεις ε, από κυβερνήσεις, ε, από ενδιαφερόμενους ε, και άλλους. Αυτό είναι μια πολύ καλή βάση για να οικοδομήσουμε την πρότασή μας για τα μελλοντικά προγράμματα τα οποία θα υπορθούν το δεύτερο εξάμεινο του 2011. Έχουμε λοιπόν σε διοικητή της νεολαίας σε δράση, οι συζητήσει και τα αποτέλεσμα συζητήσεων θα συμπεριληφθούν σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά υπάρχει ένα χωριστό χρονοδιάγραμμα, αν θέλετε, για την πρόταση, για την υποβολή κάποιων προτάσεων. Θεωρούμε λοιπόν ότι επειδή υπάρχουν όλε αυτέ τις πολιτικές δεσμεύσει σε ζητήματα κινητικότητα, ε, θα υπάρξει και η δυνατότητα να αυξηθούν η χρηματοδότηση και δεν βλέπουμε πώς θα μπορούσαμε να πετύχουμε τους στόχους αυτούς αν δεν υπάρξουν περαιτέρω κονδύλια. Και τα προγράμματά μας μέχρι τώρα ε, ε, στέφθησαν από επιτυχία. Άρα αυτό είναι ένα καλό δείγμα. Να σχολιάσω τώρα σε κάποια ζητήματα που εθίγησαν. Εκφράστηκαν ανησυχίες ε, σχετικά με αυτή την πρωτοβουλία ranking, την ε, ταξινόμηση αν θέλετε. Δεν νομίζω ότι ο όρος ranking είναι ο καλύτερος όρος για αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε. Αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι να έχουμε ένα εργαλείο φιλικό προς το χρήστη που θα βοηθάει τους ε, φοιτητέ προκειμένου να γνωρίζουν τι και πού να σπουδάσουν, αλλά να έχουμε και ε, φορείς που θα μπορούν να ε, χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο για να εξεύρουν συνεργάτες, εταίρους κλπ. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια πολύ πιο πολυδιάστατη αν θέλετε εικόνα των ε, πανεπιστημίων και των ιδρυμάτων, όχι μόνο το θέμα της έρευνας, αλλά και της διδασκαλίας, ε, πώς διεξάγεται, καινοτομίας, μεταφορά γνώσεων, το θέμα της ε, διεθνοποίησης αλλά και ε, τις περιφερειακές ε, δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα πανεπιστήμια. Αυτό θα είναι ένα εργαλείο φιλικό προς τον χρήστη και θα προσαρμόζεται στις ανάγκες του. Θα, έχουμε λοιπόν αυτούς τους πίνακες και θα βλέπετε την αποδοτικότητα ή την επίδοση, αν θέλετε, του Πανεπιστημίου. Τώρα, για το θέμα του 40%. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την ε, ανώτατη εκπαίδευση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ε, στοχεύουμε και δεν εστιάζουμε στην περιμερή ε, κατάρτιση και εκπαίδευση. Υπάρχουν διάφορες ανακοινώσεις πάνω στο ζήτημα για τη βελτίωση της ποιότητας και την προσφορά, διαθεσιμότητα για την επαγγελματική και κατάρτιση και εκπαίδευση. Επίσης χρειάζεται να γνωρίζουμε πως ε, όταν αναλύουμε τις ε, εκτιμήσεις του Σεντεφόβια το 2020 βλέπουμε ότι έχουμε 15 εκατομμύρια ε, πλέον θέσεις εργασίας υψηλού, υψηλής εξειδικευσής αλλά έχουμε και 50% εργασίες με χαμηλότερη εξειδίκευση. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τον χρόνο που μου δώσατε. Ευχαριστούμε. Αν είναι έτσι και αν δεν κάνετε πραγματικό ράγκι, προσπαθείτε να βρείτε ένα άλλο όνομα. Είναι εύκολο. Είναι εύκολο. Τότε θα σας υποστηρίξουμε πλήρως αν κάνετε αυτή την πύλη και αν χρησιμοποιήσετε άλλο όνομα δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν λέτε όμως ranking, κατά, κατάταξη σημαίνει κατάταξη και δεν μας αρέσει αυτό. Έχουμε το Εράσμου, το Κορμένους, όλα αυτά τα προγράμματα δεν χρειάζονται. Ναι, είναι αλήθεια, αλλά δεν το αναφέρετε στο πρόγραμμα εργασίας σας. Και γιατί. Πρέπει να κάνετε τη δουλειά σας, το εκτιμούμε. Αλλά δεν μας αρέσει η απάντησή σας γιατί δεν μπορούσατε να δώσετε την απάντηση που ήθελα εγώ να ακούσω γιατί δεν υπάρχει τέτοια απάντηση. Φόβο βλέπω. Μιλάμε, μιλάτε για χρήματα, για αυτά τα προγράμματα και φοβόμαστε ότι δεν θα υπάρχουν πολλά χρήματα. Αυτό είναι το πρόβλημα και νομίζω ότι αυτό είναι που κρύβεται πίσω από την ε, συμπεριφορά της Επιτροπής. Πρέπει λίγο να το αντιμετωπίσετε αυτό. Σας ευχαριστούμε για την προσπάθειά σας. Προσπαθήσατε να μας δώσετε μια ιδέα για το τι σκέφτεστε γι' αυτό. Είναι κάποιος άλλο από την Κομισιόν που θέλει να μιλήσει. Κάτι καινούργιο θα μας πείτε. Morgen, Frau Vorsitzende. Καλημέρα κυρία Προέδρε, αγαπητοί ε, βουλευτές. Εγώ είμαι από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, ε, είμαι η Σάγκες Βέστφαλς και έχω ασχοληθεί με το κομμάτι της απασχόλησης αυτής της πρωτοβουλίας ε, ε, σε συνεργασία με τους συναδέλφους σας από την Επιτροπή Απασχόλησης. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες, θα κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις για να επηρεάσω την εντύπωση που υπάρχει για αυτήν εδώ την πρωτοβουλία. Όπως είπε και η συνάδελφος, δεν είναι πρόγραμμα, είναι μία εμβληματική πρωτοβουλία η οποία θα δείξει τι ακριβώς χρειαζόμαστε ώστε να έχουμε περισσότερο ανάπτυξη και θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Είπατε ότι το πλοίο δεν έχει θάλασσα για να ε, πλεύσει. Έχουμε όμως ε, θάλασσα. Έχουμε ανθρώπους που δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Έχουμε ένα χρόνο ύφωση στην Ευρώπη ε, και έχει αυξηθεί η ανεργία. Ε, πέντε εκατομμύρια είναι οι άνεργοι στην Ευρώπη, οι νέοι. Σιγά σιγά ξαναερχόμαστε πίσω στην ανάπτυξη αλλά το θέμα είναι πόσες είναι οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν σε αυτήν την νέα περίοδο ανάπτυξης. Αλλά δεν θα είναι μια job reach recovery, μια ανά, ανάνυψη της οικονομίας που θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας. Θα είναι καλό λοιπόν ε, ε, να υπάρχει ε, αυτό το υπόβαθρο που θα βοηθήσει τους νέους να ενσωματωθούν και πάλι στην αγορά εργασίας. Ε, και αυτό είναι και το κεντρικό σύνθημα αυτής της πρωτοβουλίας της Κομισιόν, να τους βοηθήσει να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτό το μεταβατικό στάδιο ε, και να πάρουν την κατάλληλη κατάρτιση που θα τους βοηθήσει να μπουν στην αγορά εργασίας. Ας πούμε, υπάρχει μείωση των ανθρώπων που φεύγουν νωρίς από το σχολείο. Και πραγματικά όταν βλέπετε τους άνεργους, αυτά τα 5 εκατομμύρια, βλέπετε ότι αυτοί ε, στην πλειονότητά τους έχουν τέτοια προβλήματα, δεν έχουν τελειώσει π.χ. το σχολείο. Αυτό ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω. Δεν είναι ένα πρόγραμμα που θα αντικαταστήσει άλλα. Γιατί δεν υπάρχει πολιετές πρόγραμμα, ρωτήσετε. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, πολλοί κονδύλια έχουν ε, τα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τέτοια προγράμματα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε ότι δεν... το ξέρουμε ότι δεν είναι πρόγραμμα. Και θα έλαμε να εμποδίσουμε απλώς το να γίνει πρόγραμμα, να το εμποδίσουμε από το να γίνει πρόγραμμα. Δεν θέλουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί δεν αναφέρονται το Εράσμος, το Λεωνάρτο, τίποτα η λέξη εμβληματικός ε, στο υπόβαθρο δεν επαρκεί. Θέλουμε λοιπόν για άλλη μια φορά να τονίσουμε ότι αυτή η ιδέα είναι λίγο περίεργη. Ότι θα φέρουμε στα κράτη-μέλη ιδέες και γνώσεις που δεν έχουν ως τώρα. Το θέμα της απασχόλησης και της εκπαίδευσης. Καλό θα ήταν να γινόταν αυτό, αλλά το αμφισβητώ. Τώρα για τους ανθρώπους που φεύγουν νωρίς από την εργασία, είναι από το σχολείο, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να πάμε στο 15%. Από το 15% στο 10%. Για αυτούς τους ανθρώπους καλό θα είναι όχι να τους ε, βοηθήσουμε να σπουδάσουν, αλλά να κάνουν μια επαγγελματική κατάρτιση. Αυτοί δεν θα πάνε στο πανεπιστήμιο. Εμείς θα μιλάμε καλύτερα για ένα καλύτερο σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης. Παρόλο που η, η, κρίση στην ε, Γερμανία δεν ήταν ακριβώς ίδια όπως και στις άλλες χώρες, έχουμε λιγότερη απασχόληση, ε, ε, ε, ε ανεργία συγγνώμη στους νέους γιατί έχουμε χώρες με 25 και 30% ανεργία και σε εμά έχουμε μόνο 10%. Υπάρχει λόγος. Είναι ότι η επαγγελματική εκπαίδευση σε κάποιες χώρες δεν αντιμετωπίζεται σωστά και ίσως θα έπλεπε κάποιος από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει κάποια κίνητρα και κάποιες βέλτισεις πρακτικές. Αυτό δεν θα γίνει με τους νέους εν κινήσει. Ε, αυτή ήταν η τελευταία μου λέξη. Ίσως και εσείς να θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος κύριε Πρόεδρε και για να σας πω κάτι πάνω σε αυτό που εσείς μας εξηγήσατε. Όντως, σε Γερμανία και Αυστρία υπάρχει όντως αυτό το διτό σύστημα και με αυτό το σύστημα διευκολύνεται η είσοδος στην αγορά εργασίας. Ναι, αυτό είναι σωστό, γιατί υπάρχει εξάσκηση πρακτική, κατά τη διάρκεια της φίτησης, και έτσι κανείς αποκτά τις δεξιότητες που χρειάζονται. Όμως υπάρχει και άλλη μια πλευρά σε αυτό το ζήτημα. Για παράδειγμα, εάν εκπαιδεύσουμε τους νέους μόνο για τη δουλειά, μόνο για την ε, απόκτηση ειδικών δεξιοτήτων και την ε, γενικότερη εκπαίδευση την παραλείψουμε, την αγνοήσουμε, τότε αν χάσουν τη δουλειά για την οποία εκπαιδεύτηκαν, Πώ θα βρουν άλλη δουλειά, δεν θα έχουν την γενική παιδεία που χρειάζεται. Όλα χρειάζονται για να μπορεί κανεί να έχει την ισορροπία μεταξύ των ε, γενικών ικανοτήτων και των ειδικών δεξιοτήτων που απαιτούνται. Επομένως, είναι αποτελεσματικό το σύστημα αυτό που έχετε. Θα πρέπει να ξέρουμε όμως ποιες είναι οι συνέπειες από αυτή την πολιτική. 40% ξέρετε των ε, πτυχιούχων έχουν καλυφθεί από αυτήν τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Να κάτσουμε όμως και να προσθέσουμε 30% αυτών των βαθμίων. Ε, διπλωματούχων που εξήγησε κυρία Πρόεδρε. Τότε να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε. Γιατί να δούμε αν μπορούμε να φτάσουμε το 40% στι ΗΠΑ και 50% στις, ε, στην Ιαπωνία. Όμως η Ιαπωνία και είπα η επένδυση ανά φοιτητή είναι δύο-τρεις φορές πιο μεγάλη από ό,τι στην Ευρώπη. Και αυτά εξασφαλίζονται από ιδιωτικό χρήμα και κρατικό. Γι' αυτό σας λέω ότι εκεί πέρα επενδύουν περισσότερα από την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ για όσα είπατε. Εγώ θα προσπαθήσω όσο γίνεται περισσότερο να καλύψω όλα όσα είπατε και τώρα. Ναι, είναι αλήθεια ότι τώρα ξέρω τι θα πρέπει να λάβω υπόψη και δεν θέλουμε να υπάρχει αυτή η όπω τα άλλα προγράμματα. Θέλουμε όμως να εισφέρουμε κάτι καινούριο. Ε, γιατί όλοι θέλουμε ή στην Ευρώπη να εφαρμοστεί μια τέτοια στατική. Το συντομότερο δυνατόν. Γι' αυτό σα παρακαλώ να τα ξανασυζητήσουμε ε, τον Ιανουάριο. Τότε θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε όψεις εκ νέου. Θα γίνει μια δεύτερη ανταλλαγή απόψεων με την σχέδιο ε, και θα γίνει ψηφοφορία στην Επιτροπή τον Μάρτιο και στον Απρίλιο στην Ολομέλεια. Πάμε στο σημείο 11, μάθηση κατά πρώτα έτη τη ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Χάνιμπουλ έχει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αρχίζω αναφέροντά σα. ότι δεν θεωρώ ότι αυτό το οποία λέμε τώρα θα μετουσιωθούν σε πρόγραμμα στο εγγύς μέλλον. Όμως ας γίνουν μια τέτοια πρωτοβουλία. Ίσως βέβαια να μην καταλήξουμε να παρέχουμε πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες. Should start moving our attention towards and start... Να αρχίσουμε επομένω να προβληματιζόμαστε στα σοβαρά για αυτές τις εμβληματικέ πρωτοβουλίες και να δούμε τι γίνεται αυτούς που νωρίς εγκαταλείπουν το σχολείο. Μήπως και με κατάλληλε ενέργειες τα πρώτα χρόνια του σχολείου, που είναι το θεμέλιο και η βάση για τη συνέχεια, μπορέσουμε να μειώσουμε αυτούς που εγκαταλείπουν το σχολείο. Τέλος πάντων, ευτυχώ που τουλάχιστον θίγουμε τώρα το θέμα σήμερα. Δεν, περιμένω, όπως σας είπα, να έχουμε και πολλά στη συνέχεια, αλλά τουλάχιστον τώρα ε, το, το ξεκινάμε και επομένως Μόνο το θέμα τώρα φύγεται και εξετάζεται. Και όπω και για όλα τα άλλα που συζητήσαμε, για την ανωτέρα εκπαίδευση, για του νέου κλπ. Εδώ έχουμε πάλι μια πολυμορφία παραδόσεων στην Ευρώπη. Αυτό είναι αναμενόμενο. Και Επομένω, μεγάλε είναι διαφορέ στο τι παρέχεται, η ποιότητα, τι γίνεται με τι υπηρεσίε, ε, το των αρχών Επομένως, δεν είναι δυνατόν να έχουμε ενιαία προσέγγιση. Και αυτό το οποίο θα πρέπει ή το μέλλον να φροντίσουμε είναι να έχουμε κάποιο είδου πλαίσιο πανευρωπαϊκό. Κοινέ αξίε και ιδέε για το τι θέλουμε να γίνει όσον αφορά τη, τα, τα, τα, πρώτα χρόνια της ε, εκπαίδευσης. Και να δούμε τι θα προκύψει. να κάτσουμε επομένω να πάρουμε τι διαφορετικέ ρυθμίσει των μελών και να δούμε τι μπορούμε να βγάλουμε σαν κάτι το οποίο να έχει συνοχή. Γιατί βέβαια όλα τα πράγματα επιδέχονται βελτίωση, άρα και εν προκειμένου κάτι μπορεί να βελτιωθεί. Πριν μπούμε στι λεπτομέρειε, θέλω να σα πω ότι στην έκθεση θα ασχοληθώ με την ηλικία μέχρι τα 6 Καλά, αλλού βέβαια κανείς ε, θα κάνει τα ίδια 4,5-5 χρόνια, εξαρτάται. Ή καμιά φορά κανείς μπαίνει στην εκπαίδευση πιο νωρίς, αν έχει γεννηθεί πιο νωρίς. Τέλος πάντων, έχουμε αυτό το συμβούλιο που είναι στη Βαργελόνη και είπαμε να καλυφθούν τα παιδιά αυτά ε, τριών ετών και είπαμε ότι 33% των παιδιών που καλύπτονται είναι κάτω από 3. Είναι κάποιοι στόχοι που δείχνουν μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη την αγορά εργασία. Αυτό έχει οικονομική σημασία. Όμως θα πρέπει να δούμε πώς θα ωφεληθούν και τα παιδιά. Άρα διπλή προσέγγιση χρειάζεται. Τα αποτελείο για και από την άλλη μεριά τι επιπτώσεις θα υπάρχουν για αυτά τα παιδιά και τι σημασία έχουν όλα αυτά για το όταν θα μεγαλώσουν. ισότητα ευκαιριών, είχε ληφθεί υπόψη για αυτές τις εξαγγελίες της Βαρκελόνης. Δεν είναι κακά αυτά Α συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψη. απλώ θα πρέπει εμεί να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Να δούμε το ευρύτερο τοπίο για αυτή την τρυφερή ηλικία. Δηλαδή ότι η παιδική σταθμή δεν είναι ένα πάρκινγκ για παιδιά. Είναι κάτι το οποίο συμβάλλει στην ανάπτυξή τους στο μέλλον τους. Και επηρεάζει την κοινωνία σε όλη την Ευρώπη. Φυσικά και υπάρχουν οφέλη οικονομικά. Το οποίο έχει σημασία ιδίω στη σήμερα ημέρα. Έτσι όπω πάει η οικονομία. Όλα θα ληφθούν υπόψη και είναι κρίμα που όταν μιλάμε για οικονομικά ωφέλη και ωφέλη γενικότερα για αυτή την ηλικιακή ζώνη 0 έως 6 επενδύουμε λιγότερα από ότι σε άλλες φάσεις της διαδρομής της εκπαίδευσης. Επομένως, ίσως δεν υπάρχει τόσο προσβασιμότητα όσο θα έπρεπε να στον πώς υπήρχε για να δούμε τι γίνεται και με αυτό το δίκτυο για την φροντίδα των παιδιών. Ξεκινάει αυτή η ιστορία από το 1996 και είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε 1% του ΑΕΠ για αυτά τα πρώτα χρόνια, αλλά μόνο μόνο 5 χρόνια έχουν προσεγγίσει σε αυτό το στόχο. 5 από τα 27, δεν θα πω ποια κράτη είναι, αλλά λίγο είναι και μιλάμε για κάτι που έρχεται το 96, επομένως αυτό δεν είναι πάρα πολύ καλή επίδοση. Γι' αυτό σα λέω ότι ακόμα έχουμε πολλά που μα περιμένουν, που θα πρέπει να τα προσέξουμε. Έχουμε επομένω ε, όλε αυτέ τις ενδείξεις. Ότι δηλαδή ό,τι προσπάθεια γίνεται σε αυτά τα πρώτα χρόνια αποδίδει πολύ περισσότερο από οτιδήποτε γίνει σε άλλη φάση. προοπτικές απασχόλησης επίσης. Και αυτό έχει σημασία και όσον αφορά αυτούς που καταλήγουν το σχολείο νωρίς. Άρα είναι μια επένδυση στην οποία θα πρέπει να προβούμε. Μια επένδυση που θα πρέπει να πλαισιώνεται με κίνητρα. Θα πρέπει το θέμα αυτό να το δούμε καλύτερα και ευρύτερα. Δεν είναι πολυτέλεια να τα προσέξουμε αυτά που γίνεται τα πρώτα χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Όλα αυτά έχουν σημασία μεγάλη. Τέτοια προσέγγιση θα πρέπει να γίνει στο θέμα και νομίζω ότι θα βοηθήσει την Ευρώπη μακροπρόθεσμα. Αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για μακρόπνοη προοπτική, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στα σοβαρά. θα έχει επιπτώσεις οικονομικές σοβαρές στο Και λέγοντας αυτό, φυσικά, ξέρω δεν είναι αυτονόητο έτσι όπως είναι η συγκυρία οικονομική τη σήμερα ημέρα. Ξέρω όμως ότι υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για αυτή την ε, ηλικιακή ζώνη. Και, επομένως, θα πρέπει η Επιτροπή μας να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα αυτό. Για να κάτσουμε επομένως να το μελετήσουμε. Από την πλευρά του παιδιού. Να δούμε ποια είναι τα πιο σημαντικά. Ποια είναι τα προβλήματα σε αυτή την ε, τριβερή ηλικία. Έτσι να δουλέψουμε με ανοιχτό μυαλό, να λάβουμε υπόψη τις καλύτερες πρακτικές, να λάβουμε υπόψη την ακαδημαϊκή, την πανεπιστημιακή έρευνα, υπάρχει πολύ υλικό εκεί. Να το πάρουμε στα σοβαρά. Έχουμε διαπιστώσει στην Επιτροπή μας ότι τα παιδιά έχουν πολλές δυνατότητες, είναι και αυτά πολίτες, ε, ε, ενεργοί πολίτες, οι απόψεις τους έχουν σημασία. Όλα αυτά πρέπει όμως να τα μετουσιώσουμε στο πώς θα διαμορφώσουμε την παιδεία για αυτή την πρώτη φάση της ζωής τους. Την πλευρά των παιδιών να το δούμε. Τα ξέρετε, αλλά και πάλι θα σας πω ότι η περίοδος από τη γέννηση μέχρι τα τρία χρόνια είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Αποφασιστική για το πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά, ο εγκέφαλος, η η γνωστική τους ικανότητα, η γλώσσα, μαθηματικά, όλα αυτά που είναι πολύ σημαντικά για τα παιδιά και για την κοινωνία στο μέλλον. Είναι το θεμέλιο για την ισόβια παιδεία, κατάρτιση, εκπαίδευση, όλα αυτά που μας απασχολούν εδώ. στόχοι της Λισαβόνας. Άρα, καλή πλαισίωση για τα πρώτα χρόνια, όπου είναι αποφασιστικό τι παιδεία θα υπάρχει, για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας. Αυτό να ληφθεί υπόψη και να πλαισιωθούν κυρίω οι μειονεκτούσε, οι μη προνομικέ οικογένειε, γιατί αυτέ χρειάζονται πλαισίωση. Σε πολλά κράτη-μέλη, σίγουρα στη δική μου χώρα, όπου έχουμε Περισσότερα βέβαια κέντρα για πλαισίωση αυτή τη τροφιστική όπω είχαμε πριν από λίγα χρόνια. Ποιοτική ε, προσπάθεια έχει γίνει αυτή και φυσικά είναι πολύ δάπανε αυτέ οι προσπάθειε, αλλά ε, θέλουμε ε, να υπάρχει προσβασιμότητα και όλοι όσοι χρειάζονται την πλαισίωση να μπορούν να την έχουν. Η διδασκαλία είναι κάτι που σημαίνει ότι εκμάθηση συνδυάζεται με φροντίδες. Και εμείς ε, και τα κρατημέλη θα πρέπει έτσι να βλέπουν τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι έχει προσεχθεί αυτό το θέμα τόσο πολύ. Ή ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων. Υγεία, ανάπτυξη σε αυτή την τρυφερή και τόσο σημαντική ηλικία. Όλα αυτά θα πρέπει να μας αποσχολήσουν. Και να αρχίσει ο προβληματισμός και να δούμε προς τα πού θέλουμε να, πάει το πράγμα. Ανταλλαγή των αρίστων πρακτικών, μια που τα κράτη-μέλη έχουν πολλά να διδάξουν το ένα στο άλλο. Άρα κάποια στιγμή αυτή η ανταλλαγή προτάσεων αρίστων πρακτικών είναι κάτι που θα αναδείξει ως προτεραιότητα την ηλικία για την οποία συζητούμε. Και αυτό θα καλύψει και την κινητικότητα των δασκάλων, νηπιαγωγών, όλων αυτών που ασχολούνται με τα παιδιά και με την ανταλλαγή, μόνο θα μάθει από τον άλλο και θα έχουμε ένα καλύτερο πλαίσιο να κινηθούμε. Και θα φροντίσουμε τα παιδιά καλύτερα. Βέβαια, ακριβώ επειδή δεν υπάρχουν πόροι άμεσα, δεν θα υπάρχει και πρόγραμμα άμεσα, αλλά ο προβληματισμό είναι σημαντικό να μπει στη μεσή διάταξη. Να το συζητήσουμε και να κάνουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Ευχαριστούμε κυρία Χάνιμπαλ. Kiitoksia puheenjohtaja. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. ακούγοντας την κυρία Χάνιμπολ μου ήρθαν στο μυαλό μία σειρά από ζητήματα Μιλήσα, άκουσα για ανάπτυξη του γνωστικού κλπ. Υπάρχουν μία σειρά από θεωρίες ε, που υπάρχουν σχετικά με την ε, εξέλιξη των παιδιών 0 με 3, 3 με 6 και ούτω καθεξής. Συμφωνούμε ότι πρόκειται για μια ζωτική σημασία ηλικία για την ε, εκμάθηση. Όπως και να έχει αυτή η θεωρία, πιστεύω ότι το καλύτερο είναι να φροντίσουμε τα παιδιά μας ε, με αγάπη, στοργή. Αυτό είναι πολύ καλύτερο και θα επιτρέψει να ξεπεράσουμε ενδεχόμενα προβλήματα, να ξεπεράσουμε όλο το παιδί ενδεχόμενα προβλήματα διδασκαλίας, διαπαιδαγώγηση από το σχολείο κλπ. Εμείς πρέπει να θρέψουμε το, τα παιδιά μας επαναλαμβάνω με στοργή και αγάπη. Δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορούσα να εκφράσω μια φιλελεύθερη άποψη, αλλά Είμαι της γνώμης ότι χρειάζεται να έχουμε τις ε, οικουμενικές αξίες, τις ανθρώπινες αξίες που θα βρίσκονται στη βάση της, ε, της εκπαίδευσης ε, και της ανατροφής του παιδιού μας. Θα μπορούσα να πω τις χριστιανικές αξίες που προσφέρουμε στα παιδιά μας ανά πάσα στιγμή. Όταν διαβάζω αυτές τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μου δίνεται η εντύπωση πως ε, έχουμε μια αντίληψη κάπως παράδοξη της ζωής. Αλλά γεννήθηκε ένα παιδί σε μια οικογένεια και μετά όταν διαβάζουμε τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις σε ό,τι φορά το ΑΕΠ και μας ήρθε στο μυαλό η στρατηγική Λισαβόνας και η στρατηγική του 2020. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι μιλάμε για μια γένεση, κάτι το εξαιρετικό, κάτι το πολύ σημαντικό, μια νέα ζωή. Κάθε παιδί λοιπόν έχει το δικαίωμα να ζήσει μια αξιοπρεπή ζωή μέσα από την αγάπη και την στοργή των γονιών. Τα παιδιά δεν έρχονται για να προσφέρουν περισσότερο στο ΑΕΠ, έρχονται στη ζωή για να ζήσουν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να θεωρήσουμε το παιδί ως παιδί, τελεία και παύλα. Ως ανθρώπινο όν μπορείτε να μιλήσετε με οποιουσδήποτε ορισμούς, αλλά θεωρώ ότι το παιδί έχει δικαίωμα στην παιδική ηλικία. Ίσως ε, να θεωρήσουν πολύ ότι ήμουν αυστηρός απέναντι στα παιδιά μου τα πρώτα χρόνια της ε, ζωής τους, αλλά ήταν οι καλύτερες στιγμές της ζωής μου όταν παρατηρούσα τα, τα παιδιά μου να μεγαλώνουν. Εγώ πιστεύω σε ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στην αγάπη. Τώρα, ε, Ξέρετε ότι σήμερα με τα ε, σχολικά μας συστήματα τα παιδιά μαθαίνουν ανάγνωση από τα επτά τους. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αν μπορεί να γράφει, να διαβάζει στα επτά ή στα οκτώ. Εγώ αυτό που θέλω είναι το παιδί να μπορεί να παίζει, να μπορεί να παίξει, να ζήσει την παιδική του ηλικία. Αυτό φρονώ. Αυτό νομίζω ότι κάνει το μοναδικό τον χαρακτήρα της ανθρώπινης φύσης και ζωής. Πρέπει να αναρωτηθούμε πώς θα δημιουργήσουμε τις καλύτερες προϋποθέσεις ώστε οι γονείς να καταστούν οι καλύτεροι γονείς για τα παιδιά τους και να τους προσφέρουν τις μεγαλύτερες <clears throat> δυνατότητες για να ανατροφούν, ανατραφούν σωστά και να τα διαπαιδαγωγήσουν σωστά. Ε, ε, αυτά πιστεύω φαίνεται πως, ε, μάλλον σας φαίνεται πως κάνω κήρυγμα, αλλά αυτές είναι οι ιδέες μου. Πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά να αναπτυχθούν με τον καλύτερο τρόπο. Δεν χρειάζεται να είμαστε πολύ αυστηροί, να τους βάλουμε κανόνες. Αυτά θα σταματήσω για να μην σας ζαλίσω. Yeah, vielen Dank. Ευχαριστούμε. Ξεχάσατε να τραγουδήσετε τραγούδι. Συνεχίστε, μπορείτε ναι. εσείς να τραγουδήσετε. Δεν ε, θα το κάνω. Είναι δύσκολο για μένα να παρακολουθήσω αυτή τη φιλοσοφική σκέψη σήμερα το πρωί. Μάλλον θα πρέπει να πάω στη Φιλανδία μια βόλτα. Ήταν πολύ σημαντικά όλα όσα είπε η Μέρη για την σημασία αυτού του τομέα. Πρέπει στα κράτη-μέλη να τονίσουμε τη σημασία της ε, πρώιμης μάθησης και ε, πόσο, σημαντικό είναι να βάλουν τα παιδιά στο σωστό δρόμο. Δίνουμε έμφαση στις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτόν τον κλάδο λοιπόν είναι σημαντικό να γίνει το ίδιο. Πρέπει να μιλήσουμε για αγάπη, για πειθαρχία, ε, γιατί υπάρχουν πολλές οικογένειες που είναι μονογονεϊκές τα παιδιά χρειάζεται να έχουν ε, κάποιο πρότυπο στη ζωή τους ε, για να μάθουν ε, πώς να συμπεριφέρονται, πώς να είναι στη ζωή τους. Και γι' αυτό πραγματικά προσβλέπω σε μια καλή συνεργασία με την κυρία Μέρη, με τη Μέρη σε αυτό. Κύριος Μπόρης. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση του θέματος. Ευχαριστούμε και τον κύριο Τάκουλα για την ε, φιλοσοφική αντιμετώπιση του ζητήματος. Εγώ έχω παιδιά και έχω ασχοληθεί στην πράξη με το θέμα. Είναι γεγονός ότι τίποτα δεν ε, αντικαθιστά τους γονείς ε, στην ανατροφή του τέκνων τους. Εάν δεν υπάρχει αγάπη στο σπίτι και ιστορία είναι πολύ δύσκολο εκ των υστέρων να αντιμετωπιστούν ε, τα διάφορα προβλήματα και οι φραγμοί οι προκαλούνται. Και αυτή η πρόορη εκπαίδευση στην οποία αναφέρεστε θα πρέπει να λάβει υπόψη και αυτό το στοιχείο. Οι γονείς δεν προσφέρουν πάντα σε αυτήν την ε, ανατροφή στα παιδιά τώρα. Η ε, εκπαίδευση σχολική, προσχολική, πώς μπορεί να εξορπίσει τα πράγματα σε θύματα αξιών και άλλων. Πώς ε, να ε, ασχοληθούν με τα θέματα και τα προβλήματα των παιδιών, ε, χωρισμένων γονιών και όχι μόνο αυτό, από παιδιά τα οποία δεν έχουν λόγο ε, απόστασης ε, από τα σχολεία δεν έχουν δυνατότητα να πάνε σε νηπιαγωγία, δηλαδή σε μια προσχολική εκπαίδευση. Στη χώρα μου πολλά κονδύλια έχουν δοθεί για την κατασκευή νηπιαγωγείων ε, και προνηπιακών σταθμών το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ε, χρηματοδότησε ε, σημαντικά αυτές τις προσπάθειες ε, για τη μεταφορά των παιδιών κλπ. Και τα προβλήματα που ξεπεράστηκαν ε, ήταν τα παιδιά τα οποία δεν είχαν δυνατότητα να πάνε στην υπηαγωγία, στους παιδικούς σταθμούς, μπόρεσαν να φτάσουν σε αυτούς. Τους ανοίχθηκαν λοιπόν και αυτές οι πόρτες ε, και η υγιεινή βελτιώθηκε στα, για τα παιδιά στις ε, περιοχές της Υπέθρου. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα πολύ σοβαρά. Η χρηματοδότηση γίνεται και από τα κράτη-μέλη αλλά και με τη βοήθεια του χρηματοδοτικού του κοινωνικού ταμείου. Κάτι άλλο το οποίο πρέπει να μας προσχολήσει είναι η οικογένεια. Συχνά αυτή η ανατροφή, αυτή η εκπαίδευση που γίνεται πριν από την έναρξη ε, σχολικού βίου είναι ένα θέμα στο οποίο εμπλέκονται ιδιαίτερα οι μανάδες και πολλές φορές ε, όταν υπάρχουν προβλήματα στις οικογένειες αυτό ε, οφείλεται και σε ζήτημα αγοράς εργασίας ε, υπάρχει, διότι υπάρχει ο αποκλεισμός ε, κάποιων γονιών από τον χώρο της εργασίας κλπ. Κύριε Φεχάνη, ευχαριστώ. ακούσαμε πολλά για την αγορά εργασία για τους ανθρώπους που βγαίνουν από αυτή. Μιλήσαμε για την οικονομική σημασία για τη, της ε, εκπαίδευσης. Ο κύριος Τακούλα ανέφερε πιο ηθικές, πιο, κάποιες πιο ηθικές και φιλοσοφικές διαστάσεις. Γενικά το σημαντικό είναι να αναθρέψουμε τα παιδιά μας με τέτοιο τρόπο και να τους δώσουμε τις σωστές ε, ε, τεχνικές. Ο κύριος Στακούλα είπε ότι έζησε πέντε ε, πολύ εντατικά χρόνια. Έχει λοιπόν κάποια γνώση. Από τη στιγμή που τα παιδιά κάθονται μπροστά στην τηλεόραση και βλέπουν το τελετάπης και τέτοια είναι η ανατροφή που παίρνουν στην οικογένεια, μάλλον πρέπει να σκεφτούμε ποιες είναι οι ευκαιρίες που έχουν τα παιδιά. Και για μένα δεν είναι το θέμα εάν η γυναίκα θα γυρίσει γρήγορα στη δουλειά ή όχι, αλλά πώς ε, θα μπορέσει ε, το παιδί να έχει την οικογένειά του στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Νομίζω ότι αυτό είναι και η αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ε, θα πρέπει αυτά να φροντίσουν. Θα πρέπει να μπορέσουμε μια ολόκληρη γενιά να τη διαμορφώσουμε έτσι, να βοηθήσουμε τις γυναίκες με την αγορά εργασίας, γιατί η αγορά εργασίας χρειάζεται τις γυναίκες, χρειάζεται εξειδικευμένες, ε, εξειδικευμένους απασχολούμενους. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια εναλλακτική λύση, όχι είτε αυτό είτε εκείνο. Θα πρέπει να δούμε πώς ε, θα δώσουμε τις γονείς ε, ικανότητες ανατροφής, ε, πώς θα δώσουμε στην οικογένεια τη διάσταση που πρέπει, γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία ε, πάνε στο νηπιαγωγείο και στο σχολείο από πάρα πολύ νωρίς και δεν έχουν και σωστά πρότυπα. αν υπάρχει λοιπόν μια βέλτιστη πρακτική ε, καλό θα είναι να την ξέρουμε, αλλά ένα πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο λίγο δύσκολο μου φαίνεται. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι διαφορετικές ε, οι ανάγκες και οι στόχοι και θα πρέπει αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας. Η μάθηση κατά τα πρώτα έτη της ζωής, ε, στον υπηαγωγείο, στο βρεφονιπιακό σταθμό, είναι με ένα θέμα, αλλά και εμείς ως γονείς θα πρέπει να έχουμε τις κατάλληλες δεξιότητες. Η ποιότητα επίσης της φύλαξης των παιδιών είναι σημαντική. Όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Είναι διαφορετικές οι ανάγκες. Το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει διαφορετικά να τα αντιμετωπίσει. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάνιμπαλ είπε συγκεκριμένα ότι δεν θέλει να γίνει πρόγραμμα, αλλά να γίνει ευαισθητοποίηση για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα, μένουν πέντε χρόνια στο σπίτι με τα παιδιά και να έχουν μια γυναίκα ή έναν άντρα που θα βγει για να βγάλει τα προς το ζήν. Ίσως οι γονεί ε, δίνουν πολύ περισσότερα στα παιδιά από ό,τι θα μάθαιναν στο σχολείο και στο βρυφανιπιακό και το νηπιαγωγείο. Και σε πολλές οικογένειες ακόμα ε, αυτή τη στιγμή ευτυχώς ε, υπάρχει δυνατότητα να μείνουν οι γονείς στο σπίτι, όμως σε άλλους δεν γίνεται. Και από τη στιγμή που υπάρχουν κάποιες βέλτιστες πρακτικές, είναι καλό να δοθούν ως ε, πρότυπο και όταν γίνει μια συζήτηση σε επίπεδο υπουργών, καλό θα είναι να παρουσιαστούν. Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τους ανθρώπους που φεύγουν νωρίς από το σχολείο, για τα παιδιά που δεν τελειώνουν το σχολείο, για το προγράμματα φοιτησης. Εμείς απλώς αναφέρουμε κάποια πράγματα σε σχέση με τα πρώτα έτη της ζωής. Εγώ είμαι γιαγιά, ήμουνα και μαμά και ξέρω πραγματικά ότι όλα τα μαθαίνουν τα παιδιά όταν είναι μικρά. Θα, θα, πάθ, θα μάθουν όλο και περισσότερα, θα μάθουν όσα τους δώσουμε εμείς. Όσο περισσότερα τους δώσουμε, τόσο πιο πολλά θα μάθουν. Υποστηρίζω λοιπόν την κυρία Χάνιμπαλ στην έκθεση πρωτοβουλίας. Ε, ο Άνταμ Πορκόνη από την Κομισιόν θέλει κάτι να πει. Παρακαλώ, Άνταμ. Έχεις κάτι καινούριο να θα σας δείξω τι έχω. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ναι, και εμείς χαιρετίζουμε με ενθουσιασμό αυτή την πρωτοβουλία που ήρθε τη σωστή στιγμή, γιατί αν δείτε ακριβώς τι λέει στις λεπτομέρειες της αυτή η ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, του χρόνου πρόκειται να προσφιάσει μια νέα ανακοίνωση για το θέμα αυτό του χρόνου και όπως είπε και η κυρία Χάνιμπολ η κεντρική μας ιδέα είναι το να ξεκινήσει μια προβληματική ούτω ώστε να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε την διαδικασία της ε, εκμάθησης και το πώς θα μαθαίνει τον εκάτος μας από το άλλο και όπως είπαν πολλοί πολεματολόγοι αυτό είναι πάρα πολύ βασικό είναι θέμα επικουρικότητας, δεν είναι θέμα κοινωτικό. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε εδώ πέρα τις πρακτικές, αλλά δεν τις έχουμε παντού. Άρα θα πρέπει να μάθει ένας από τον άλλο και όπως τόνισαν διάφοροι, πρόκειται για κάτι που είναι καθοριστικό για όλη τη ζωή κάποιου προσώπου. Και επομένω η επέμβαση, η παρέμβαση σε αυτή τη φάση τη ζωή τη γέννηση μέχρι τα 6 χρόνια είναι πάρα πολύ βασικό. Επίση έτσι σπάμε και το, το, το φαύλο κύκλο τη ε, φτώχεια, ε, καταπολεμούμε την εγκατάλειψη του σχολείου νωρί. Και αυτό επομένως σημαίνει ποιότητα ζωής. Μόνο όμως εάν οι σχετικές παρεμβάσεις είναι ποιοτικέ το οποίο σημαίνει δόκιμες. Και δηλαδή να μην έχουν σχολική πειθαρχία από τη γέννησή τους τα παιδιά. Πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι να καλυφθεί, το πόσο σημαντικό είναι το να συνεργάζεται κανείς με τους ε, γονείς και άρα είναι κοινή πορεία μεταξύ του ιδρύματος ας πούμε και του παιδιού και όχι οι γονεί να παραδίδουν τα παιδιά στο Ίδρυμα και να μην ασχολούνται. Τα είπε κύριε Χάνιμπολ, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι σήμερα το, το αντιμετώπιζε αυτό στα θέμα απασχόλησης, να, πάνε, να είναι ελεύθερε γυναίκε να γυρίσουν στη δουλειά, αλλά από το 2006 άρχισε να ασχολείται στο θέμα της ποιότητα η, το, το Συμβούλιο, τι γίνεται με αυτό το σύστημα για την αρχή της παιδικής ηλικίας, ε, και το 2009 συμφωνήθηκαν οι προτεραιότητες. Συντονισμός, παιδεία σε αυτά τα τέσσερα χρόνια. Οπότε θα ξεκινήσουμε με την ανακοίνωση αυτή του χρόνου και επομένως ε, μας βοηθάτε πάρα πολύ με την πρωτοβουλία σας. ανοιχτή το συντονισμό. Θεωρούμε ότι θα ωφελήσει όλες τις πλευρές. Επίσης, ε, αυτό έγινε και όσον αφορά την διαβιοκατάρτιση. Και η κινητικότητα δίνει ευκαιρίες. Έχουμε το πρόγραμμα Ριάν για αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις και την κινητικότητα όλα αυτά με τη νέα γενιά προγραμμάτων πρόκειται να αναβαθμιστούν. Επίσης, πρέπει να σας αναφέρω ότι και η Ουγγρική Προεδρία που ξεκινάει τον Ιανουάριο θα το θεωρήσει θέμα προτεραιότητας. Το Συμβούλιο θα κρίνει, θα συζητήσει το θέμα και θα εκδώσει κάποια συμπεράσματα τον Μάιο. πρόεδρος. Το Comenius ρέγγιο είναι ένα πλαίσιο όπου μπορούμε να αναπτύξουμε κινητικότητα για τους διδάσκοντες και έτσι οι δάσκαλοι μπορούν να πάνε από τον ένα στο άλλο και να ανταλλάσσουν τις καλύτερες των πρακτικών. Χάνο, θες να τραγουδήσεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ναι, αλλά μόνο οι δυο μας. Θα στο αφιερώσω. Ε, νομίζω ότι το ουσιώδες είναι να μην χάσουμε την εστίαση τη σωστή που πρέπει να δώσουμε. Ίσως ε, να μην έδωσα τα κατάλληλα παραδείγματα. Ναι, εγώ τραγουδούσα, τραγουδούσα και στο σπίτι. Α, εντάξει, θα αφήσουμε κατά μέρο όμω το θέμα αυτό. Εδώ βρισκόμαστε ενώπιον ε, ατομικών ε, αποφάσεων. Φυσικά πρέπει να λάβουμε υπόψη των ε, συμφιλίων μεταξύ επαγγελματικού βίου και οικογενειακή ζωής, αλλά υπάρχει μία τάση να εστιάζουμε στην οικονομική ζωή, στις αγορές, χρηματαγορές κλπ πρέπει ο καθένας να είναι ελεύθερος, να επιλέγει, δεν πρέπει να είμαστε συνεχώς υποχρεωμένοι να τρέχουμε πίσω από την εργασία, πίσω από τα χρήμα, το χρήμα. Αυτό ήθελα να πω. Διότι συχνά μιλάμε για την στρατηγική τη αγώνα και δεν ξέρω τι άλλο. nicht ε, ε, Ευχαριστώ. Συμφωνώ πλήρως με τον κύριο Τακούλα. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει αυτό να είναι υποχρεωτικό. Όσον αφορά στη, τα πρώτα έτη της ζωής, ε, η προσχολική αυτή πρόβλεψη θα πρέπει να είναι επιλογή για όσους τη θέλουν. Δεν έχω καμία πρόθεση να γίνει αυτό υποχρεωτικό. Έχεις ε, δίκιο, Χάνου. Τα παιδιά είναι μοναδικά. Το καθένα έχει τη δική του ζωή και προσωπικότητα. Πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι όλα τα παιδιά έχουν τις καλύτερες ευκαιρίες. Είναι λοιπόν πολύ καλό που εμείς ε, αναλαμβάνουμε αυτή τη δράση την ίδια στιγμή που η Κομισιόν θα κάνει την ανακοίνωση και η Ουγγρική Προεδρία θα το θέσει αυτό ως προτεραιότητα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πάει πολύ καλά αυτό το θέμα. Είτε στις 21 Ιανουαρίου είτε στις 3 Μαρτίου θα έχουμε την έκθεση. Θα δούμε τι θα γίνει και με την Κομισιόν. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ερχόμαστε στην πολιτική για το ραδιοφάσμα πρώτη ανταλλαγή απόψεων για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Πιστέψτε με, έχει μεγάλο υπόβαθρο στον πολιτισμό. Κυρία Καμερέβερτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχω ακούσει για τους νέους ε, την εκπαίδευση και την κατάρτιση για δύο μέρες και τώρα ερχόμαστε σε ένα πολύ τεχνικό όπως φαίνεται θέμα, αλλά όπως είπε η κυρία Πάκ, έχει και αυτό πολιτιστική σημασία πολύ μεγάλη και νομίζω ότι είναι σωστό και σημαντικό ως Επιτροπή Πολιτισμού να έχουμε μια θέση σε αυτό το θέμα του ραδιοφάσματος γιατί έχει μια πολιτιστική διάσταση και η Ήτρε που είναι υπεύθυνη επί της ουσίας θα πρέπει να πιστεί να λάβει υπόψη της και αυτά τα στοιχεία στη δική της ε, έκθεση για να διαμορφώσει την έκθεση της Κομισιόν και να την βελτιώσει προς αυτή την κατεύθυνση. Την προπροηγούμενη εβδομάδα έγινε μια συζήτηση με την Επίτροπο γι' αυτό έγινε ε, μια συζήτηση επί των σημαντικών ε, θεμάτων για αυτό το θέμα του ραδιοφάσματος. Το πρώτο στο οποίο θα πρέπει να επιμείνουμε είναι ότι πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα ε, για το ραδιοφάσμα στο οποίο πρέπει να βασιστεί στις τηλεπικοινωνίες και το πακέτο για αυτές και δεν θα πρέπει να υποσκάψουμε αυτά που μπορέσαμε να πετύχουμε με το πακέτο ε, των κοινωνιών. Σε εκείνο αναφέρεται ότι κάθε διαχείριση φάσματος πολιτιστική, κοινωνική και πολιτιστική ε, πρέπει να ε, έχει μια τέτοια διάσταση που πρέπει να υποστηρίζεται με μέτρα. Υπάρχει και την οικονομική διάσταση η οποία πρέπει να τονίζεται και εκεί ε, αναφερθήκαμε πολλές φορές στο πακέτο των τελεπικοινωνιών. Υπάρχει όμως και ένα πολιτιστικό κομμάτι το οποίο παραγνωρίστηκε. το πακέτο τηλεπικοινωνιών ε, τότε ο κύριος Μανούλα είπε ότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο που δίνονται τα, οι συχνότητες ε, έτσι ώστε να μπορούν όλοι να χρησιμοποιούν ε, προς όφελος τους αυτές τις ε, δυνατότητες. Εμείς λοιπόν τώρα θέλουμε να δώσουμε ψηφιακές δυνατότητες ραδιοφάσματος. Υπάρχουν πολλοί φόβοι όταν κοιτάζω αυτή την πρόταση της Κομισιόν που έχει κατατεθεί στο τραπέζι Έχουμε ας πούμε στη Γερμανία 800 ε, συχνότητες και πρέπει να συζητήσουμε και να δούμε τα Μεγαχέρτς και πρέπει να δούμε ότι υπάρχει και οικονομική διάσταση έτσι ώστε να, γίνει η μετα... να γίνεται η μετάδοση με τέτοιο τρόπο ώστε ο πολιτισμός ε, και η πολυφωνία στην Ευρώπη να διασφαλίζονται. Το πρόγραμμα λοιπόν για τις συχνότητες έχουν ε, και κάποιες... έχει κάποιες πολιτικές ε, διαστάσεις. Υπάρχει η ψηφιακή ε, τηλεόραση, για τηλεόραση. Ε, πρέπει λοιπόν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να σκεφτούμε ε, πώς ε, θα δοθούν οι συχνότητες, αν θα πάρουμε τις συχνότητες από συγκεκριμένους ε, που τις κατέχουν. Έτσι λοιπόν η πολιτική εδώ έχει ευθύνη. Από τη μία μπορεί να μας λένε έχουμε ψηφιακή επίγεια ραδιοφωνία ε, η Κομισιόν και από την άλλη να μας λένε ότι δεν γίνεται γιατί ε, δεν διασφαλίζεται η κινητικότητα. Το άρθρο ε, λοιπόν θα πρέπει να αναφέρεται και το πεδίο εφαρμογή και οι στόχοι πώς ακριβώς θα γίνουν όλα αυτά, πώς θα συσχετιστούν με το πακέτο ε, των τηλεπικοινωνιών, ε, πώς θα διασφαλιστεί η νομική διάσταση πώς ε, θα χρησιμοποιούνται για το δημόσιο καλό οι συχνότητες για τον πολιτισμό, για την οικονομία, επίσης για τη διαχείριση των συχνοτήτων. Όλα αυτά είναι θέματα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Η ευρυζωνική διάσταση επίσης είναι σημαντική και εδώ πρέπει σε συνεργασία με την ε, ε, Κομισιόν ε, να εξετάσουμε το θέμα της κινητής ευρυζωνικότητας. Είναι ένα θέμα που θα πρέπει να ερευνήσουμε με έξυπνο τρόπο έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τα τεχνικά και οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν δεν αναφέρεται ε, καν ακόμα αν μπορούμε μέσα από την τεχνολογία να έχουμε μια καλή μετάδοση ε, οπτικοακουστική για το DVD, DVDs, ε, πώς αυτά θα χρησιμοποιηθούν. Νομίζω ότι δεν έχει ακόμα η έρευνα ε, τελειώσει για τα 800 MHz. Στη Γερμανία έχει γίνει ε, ο διαγωνισμός, ε, δεν ξέρουμε όμως ακόμα πώς θα χρησιμοποιηθούν όλα αυτά και θα πρέπει σε επίπεδο ίντερνετ και βριζονικότητας να δούμε πώς θα λειτουργήσουν αυτά. Οι συχνότητες, όπως, είπα, όπως λέω πάντα, είναι το ψηφιακό μέρισμα το οποίο δίνεται. Οι συχνότητες είναι ένα κοινό αγαθό, πρέπει να διασφαλίζονται. Είναι και πολιτική υποχρέωση να μην χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένες επιχειρήσεις με λανθασμένο τρόπο, να χρησιμοποιούνται ε, με σωστό τρόπο και όχι να θεωρούν ότι τις έχουν και δεν θα μπορεί κανείς να τους πάρει τη συχνότητα. Επίσης για τους ε, διαγωνισμούς υπάρχει μια μεγάλη ιστορία και έχουμε δει ότι στο παρελθόν έχουν γίνει πολλά λάθη τα οποία δεν πρέπει να επαναληφθούν. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε όταν δίνουμε τις συχνότητες ε, να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούνται και σωστά και αποδοτικά. Αν είναι κάποιος άλλος που μπορεί να τις χρησιμοποιήσει καλύτερα ε, από ότι αυτόν που ήδη τις έχει να δίνεται σε αυτόν. Επίσης, και τις ε, παρεμβολές πρέπει να μειωθούν όσο γίνεται. Επίσης, πρέπει να υπάρξουν αντισταθμιστικά ε, μέτρα για αυτές τις παρεμβάσεις, ε, παρεμβολές συγγνώμη, σε συγκεκριμένες συχνότητες. Επίσης, τα σύρματα μικρόφωνα και την προβληματική με αυτά τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές αφορά τους πάντες, τη ραδιοφωνία και αυτοί δουλεύουν με αυτά και έχουν γίνει πολλές έρευνες και πρέπει λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση να έχουμε αντισταθμιστικές ε, υπηρεσίες οι οποίες ε, είναι απαραίτητες ε, σε αυτή την περίπτωση στην Γερμανία. Έχουμε εμπειρία με τα 800 MHz, μάθαμε πολλά από αυτή. Ε, όσοι, όσοι διοργάνωναν ε, ραδιοφωνικές ε, οργανώσεις, εκεί χρησιμοποιούσαν αυτά τα σύρματα μικρόφωνα. Αυτοί λοιπόν ε, συζήτησαν μαζί μας και για το κόστος δεν υπήρχε καμία ιδέα ποιος θα το επομιστεί τελικά. Είναι σημαντικό λοιπόν ε, να υπάρχουν αυτές οι αντισταθμίσεις. Ένα σχεδιασμός λοιπόν ε, σε συχνοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο μάλλον είναι κάτι που δεν θα πρέπει να γίνει, πρέπει να το αρνηθούμε. Αυτό το είχαμε ήδη συζητήσει στο ε, πακέτο των Ολυμπικοινωνιών, στο Ινωτιολογική Σκέψη 5. Να είναι αυτό στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και πάλι. Αυτό σημαίνει ότι η Κομισιόν εδώ έχει πολύ σημαντική ευθύνη, την ευθύνη να ε, πείσει τα κράτη-μέλη να διαχειριστούν σωστά τα ε, συχνότητες και να υπάρχει και συμφωνία μεταξύ αυτού και του πακέτου των τηλεπικοινωνιών, να μην μιλάνε διαφορετική γλώσσα, να είναι τα κράτη-μέλη υπεύθυνα ε, στην επικράτειά τους ε, για τις ραδιοσυχνότητες κτλ. Αυτό είναι σημαντικό να γίνει σωστά, γιατί υπάρχουν περιφερειακές και τοπικές διαφο... Ε, ιδιαιτερότητες και τα κράτη-μέλη είναι αυτά που θα πρέπει σωστά να, ελέγχουν ε, αν χρησιμοποιούνται σωστά οι ραδιοσυχνότητες κτλ. Ε, νομίζω λοιπόν ότι η Κομισιόν δεν πρέπει να αφήσει μόνο τους ε, τα ε, κράτη-μέλη σε αυτό. Θα ήταν καλό λοιπόν αν η Κομισιόν έπαιρνε κάποια μέτρα έτσι ώστε να ενισχυθεί μια συνεργασία μεταξύ των ε, κρατών μελών ε, να είναι μάλλον προμηθής η Επιτροπή σε αυτό. Και μια τελευταία παρατήρηση για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Είναι υπεύθυνη η Κομισιόν. Μάλλον εδώ είμαι λίγο έχω κάποιο σκεπτικισμό. Τι ακριβώς εννοούμε με, ε, τέτοι, με διεθνείς διαπραγματεύσεις. Τι είναι παγκόσμιες διαπραγματεύσεις για όλες τις συχνότητες στον κόσμο. Γιατί και εκεί δεν θεωρώ ότι η Κομισιόν έχει κάποιο νόημα ή έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει 27 κράτη-μέλη να διαπραγματευτούν συχνότητες σε παγκόσμιο επίπεδο θα ήταν μάλλον λογικό να διαπραγματευτεί μόνο, να διαπραγματευτεί μόνο σε επίπεδο ε, στοχοθεσίας. Αυτό θα ήταν το λογικό για μένα. Η στοχοθεσία λοιπόν ε, στη θέση μου αναφέρεται πολύ, πολύ ξεκάθαρα. Ε, μιλάω ε, για, το, για την πολιτισμική διάσταση, για τις συχνότητες, ε, συνδέω το θέμα με το πακέτο των τηλεπικοινωνιών, με τη ραδιοφωνία, γιατί θεωρώ ότι όλα αυτά είναι ένα βασικό αγαθό που βοηθά στην πολυφωνία των μέσων και που διασφαλίζει ε, αυτή την πολυφωνία στην Ευρώπη. Οι συχνότητες χρησιμοποιούνται γι' αυτό το λόγο. Δεν είναι ένα σύστημα ιδιοκτησίας ε, στην Ευρώπη όπως ε, τώρα ενδεχομένως θεωρείται και γι' αυτό αξίζει κανείς να παλέψει γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτρια. Ήσασταν πολύ αναλυτική, αλλά αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή κάποια εμπειρία, θα πρέπει να την πούμε με το όνομά της. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ των πολιτιστικών, κοινωνικών και οικονομικών πτυχών αυτού του θέματος ε, και τα πολιτισμικά θέματα, πολιτιστικά θέματα πραγματικά εδώ παραγνωρίζονται. Πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να δώσουμε και τη δική μας ε, υπογραφή σε αυτό το θέμα. το αν θα μπορούν ε, τα ε, θέατρά μας να συνεχίσουν να δουλεύουν ή να γίνονται συναυλίες. Ε, αυτά έχουν πάντοτε να κάνουν και με τις συχνότητες και το συζητάμε με την Κομισιόν γιατί μας αφορά από κοινού. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε και στους ε, συναδέλφους ότι η Επίτροπος σε αυτή την περίπτωση κάνει ακριβώς αυτό που ε, είναι προς συμφέρον των ε, πολιτών και των κρατών μελών. Κυρία Φεράνη, ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή της Πέτρα, η οποία ήταν πολύ ε, αναλυτική και έδειξε και τα βασικά σημεία αυτού του θέματος. Νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε αυτά τα, ε, αυτή την πολιτιστική διάσταση του θέματος και την κοινωνική του διάσταση και να τα δούμε πώς συνδέονται με την οικονομική διάσταση. Δεν ε, γίνεται αυτό συνήθως να ε, συνήθως ε, κοιτάμε το οικονομικό θέμα και όλοι οι άλλοι τομείς ε, παραγνωρίζονται. Πρέπει λοιπόν εδώ με τον τρόπο που αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται από την Κομισιόν που είναι μοναδικός να δούμε πώς θα δώσουμε και το στίγμα του πολιτισμού που δεν λαμβάνεται υπόψη. Η Πέτρα το ανέφερε ήδη πώς ε, θα, γίνει, ε, πώς ε, θα δοθούν αντισταθμιστικά μέτρα, πώς ακριβώς θα ποσοτικοποιηθούν όλα αυτά. Ίσως να υπάρχει κάποιο κονδύλι ένα, αλλά δεν υπάρχει ακόμα ιδέα, καμία ιδέα σχετικά με το πόσο μεγάλο θα είναι. Χρειάζεται ο κόσμος τις συχνότητες για να υπάρχουν καλύτερες επιλογές και δυνατότητες ακόμα και για τις μοιαστικές περιοχές για να μπορεί κανείς ε, να παίρνει πληροφορίες, ε, να, βοηθεί, να βοηθά ανθρώπους ε, σε επίπεδο πληροφοριών, αλλά και αρχιτέκτονες, μηχανικούς, όλα αυτά όταν μιλάμε για το φάσμα, το ραδιοφάσμα, δεν είναι ένα ξερό θέμα, έχει πολλές πτυχές και όλα αυτά περιλαμβάνονται σε αυτό. Όταν ε, ε, έχω ένα συγκεκριμένο κομμάτι του φάσματος που είναι ελεύθερο, θέλω να πετύχω κάποια πράγματα με αυτό. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε τι είναι αυτό. Θεωρώ λοιπόν σημαντικό να, να δώσουμε νέες επιλογές και δυνατότητες ε, που θα είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν, να δούμε πώς θα υπάρχει ισότητα και ένα σύγχρονος τρόπος πληροφόρησης. Και ε, αυτά που είπε η Πέτρα ε, είναι αυτό που είπε η Πέτρα είναι ότι χρειάζεται να κάνουμε και άλλα βήματα τα οποία ε, δεν είναι μόνο τεχνικά, είναι και πολιτιστικά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τρούπελ. Και εγώ από την πλευρά μου να σας ευχαριστήσω για όλα όσα είπατε. Ευχαριστώ και την και την Ζαμπίνα. Να πω στους εκπροσώπους της Κομισιόν ότι είχα συμμετάσχει ως σχεδόν στο πακέτο των τηλεπικοινωνιών και δεν θέλουμε ε, επειδή ήταν το, το τέλος της ε, περίοδου της θητείας ε, να γίνουν όλα γρήγορα. Υπάρχει μια βάση εργασίας που πρέπει να ξεκαθαριστεί όπως και τα κονδύλια. Είναι λοιπόν σημαντικό να έχουμε τη σωστή ε, μέθοδο εργασίας γιατί το θέμα του φάσματος ε, και του ραδιοφάσματος και της επίγειας ψηφιακής ε, τηλεόρασης ναι μεν παρουσιάζεται αλλά δεν βλέπουμε τους κινδύνους που έχει. Έχουμε μια εσωτερική αγορά με ψηφιακή επίγεια τηλεόραση η οποία είναι κοινή θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πολιτικές και οι τεχνολογικές επιπτώσεις αυτής. Τώρα για την πολυφωνία. Όσον αφορά στην τηλεόραση, εδώ και δεκαετίες υπάρχει ρύθμιση για την ε, πολιτισμικότητα και την πολυφωνία. Αυτή τη στιγμή σε αυτούς ε, που, στους εταιρείε κινητής τηλεφωνίας ε, που δίνουν και ίντερνετ ε, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει προστασία ειδικότερα για την πειρατεία. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε να μην δώσουμε όσο πιο πολλές συχνότητες γίνεται και να αφήσουμε ελεύθερα τα πράγματα χωρίς να υπάρχει κάποια ρύθμιση. Υπάρχουν επίσης και κάποιες σκέψεις ε, παράλληλα με την πολιτική των συχνοτήτων ε, να μην γίνουν πράγματα που τελικά δεν θέλουμε τουλάχιστον στο γραπτό κείμενο αναφέρονται κάποιες ε, πτυχές ε, ε, που μας δημιουργούν κάποιες σκέψεις. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει το θέμα και θα φροντίσει η δική μας Επιτροπή να κρατήσει μια παρουσία στο θέμα αυτό που μας αφορά πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα είπατε. Ήσασταν πολύ συγκεκριμένοι. Περιμένουμε από την Πέτρα Κάμερεβερτ την έκθεσή της. Ο συνάδελφος ε, θα μας βοηθήσει τον Απρίλιο να εγκρίνουμε την έκθεση. ο κύριος Χέκματ που κοιτάει πιο πολύ την οικονομική διάσταση, ίσως έχει κάποια δική του συμβολή και ελπίζουμε ότι τον Γενάρη θα έχουμε την πρώτη έκθεση έτσι ώστε να δούμε ποια είναι και τα πολιτιστικά στοιχεία αυτής της έκθεσης. Ευχαριστούμε πολύ. Αχ, συγγνώμη, η Επιτροπή την ξέχασα. Είναι τόσο σημαντική, παρακαλώ. Ο κύριο Οντόναλ. Looks like Irish. No? Ιρλανδικό μου ακούγεται. Α, όχι, όχι. Thank you very much, Madam Chairperson, and uh, it's very... Πολύ ενδιαφέρον συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, και να συνεχίσουμε. Εκεί που σταμάτησε η κυρία Κρούς, πριν από λίγο καιρό που ήρθε να σας μιλήσει για το ίδιο θέμα, είναι κάπως απογοητευτικό να ακούμε αυτούς τους ειλικρινούς φόβους της Επιτροπής δική σα σας στο παρελθόν που δεν τους διασκεδάσαμε. Ιδίω όσον αφορά το πόσο τώρα ε, τονίζουμε αυτό που σας απασχολεί στο πρόγραμμά μας. Γιατί δεν τονίζουμε την οικονομική πτυχή, αλλά την πτυχή της αποτελεσματικότητας. Μια από αυτό το οποίο θέλουμε είναι το φάσμα να την χάνει διαχείριση αποτελεσματικής με την ισχύουσα νομοθεσία. Αναφερθήκατε στην πέμπτη τελική παράγραφο, αλλά στην πρώτη ήδη έχουμε πει ότι αυτή η πρόταση δεν φύγει αυτή την λεπτή ισορροπία της αναθεώρησης του νομικού πλαισίου. Εμείς μόνο και μόνο θα αποφασίσουμε. Κύριε Κρούς, ήταν κρυστάλλινη πάνω σε αυτό. Επίσης, δεν υπονομεύουμε αυτήν την ισορροπία για όλα. Και για την ψηφιακή τηλεόραση σε περιφερειακό, τοπικό, εθνικό επίπεδο. Το 800 kHz αφορούν ένα κομμάτι μόνο του φάσματος. Το υπόλοιπο είναι για την τηλεόραση και δεν, δεν θέλουμε να πειράξουμε μας τις συγχρονότητες. Επίσης, αυτά που είπατε τα καλύπτουμε την πρόταση. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε πώς μπορεί να τροποποιηθεί η ρύθμιση των εκπομπών και των μεταδόσεων και να δούμε τι μεγαλύτερε αλλαγέ μπορεί να γίνουν στον αφορά τη χρήση των συχνοτήτων. Αλλά αυτό γίνεται μόνο εάν η συχνότητα χρησιμοποιηθεί από τους operators για κοινωνικού και για οικονομικού σκοπούς. Αυτό που του δόθηκε, το κομμάτι του φάσματο. Κάτι που επίσης η κυρία Κρού θέλει να είναι ξεκάθαρο είναι ότι η επίγεια τηλεόραση θα συνεχίσει όπως αποφασίζουν τα κράτη-μέλη, αλλά δεν θέλουμε να έχουμε τον κίνδυνο του να γίνει υποκατάσταση αυτής της επίγειας ε, εκπομπής με την κινητή μετάδοση. Γιατί η ταχύτητας ταχύτητα ευρυζωνικότητα είναι μια φετηρία για ανάπτυξη μιας πολιτιστικής πολιτικής σε σχέση και με την τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας. Άρα θα πρέπει οι σταθμοί να προχωρήσουν και να αποφασίσουν. Αλλά όμως αυτό θα γίνει επί τη βάση των τεχνολογικών εξελίξεων. Και θέλουν να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες ευρωζωνικότητας για να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους παντού. Τώρα, ακούσαμε πάρα πολύ προσεκτικά τι είπατε. Ήδη έχουμε αρχίσει επαφές με τους θυγόμενους και για την ψηφιακή τηλεόραση. Θα πρέπει να λέμε υπόψη ότι είναι κάτι το θετικό για τη τηλεόραση. Και τα μικρόφωνα τα σύρματα μικρόφωνα Επομένως, είναι κάτι που μας απασχολεί, έχουμε τους κατασκευαστές και όσον αφορά τα 800, τη συγγνώμη των 800, ε, εξετάζεται και θα υπάρξουν εξελίξεις σε σχέση με τις ψηφιακές εκπομπές, ούτως ώστε να δουν τα κράτη-μέλη ποια θα είναι η πιο σωστή αντιστάθμιση και η βιομηχανία να λάβει υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας. Ήδη ασχολούμεθα με αυτό, αλλά βεβαίως σωστά και προσματίζεστε για την πολυσταγική κληρονομιά. Και εμείς δεν μπορούμε να πούμε στα κατεμέλη μελη θα, πώς θα ε, χρησιμοποιήσουν τα έσοδα από τη διαχείριση του φάσματος. Πάντως, εάν θέλουν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτά τα έσοδα για αυτούς που έχουν φυγεί από την εξέλιξη για να μεταβούν στη νέα φάση και να συνεχίσουν την παροχή των υπηρεσιών. Ήδη ε, έχουμε σε επαφή με κάποιους από εσάς και θα συνεχιστεί η συνεννόηση. Πρόεδρος. Μια σύντομη πρόταση σε αυτά που μόλις είπατε. Εμείς ε, έχουμε το πρόβλημα ότι δεν βλέπουμε στο κείμενο αυτά που λέμε. Θέλουμε να σας ε, παρακαλέσουμε λοιπόν από την πλευρά της Κομισιόν να συνεργαστείτε με μας έτσι ώστε στο κείμενο να, να παραλείψουμε τέτοιες ε, τέτοια προβλήματα και κατανόησης, γιατί ε, θέλουμε ξεκάθαρα να, φέρον, να φαίνονται και οι πολιτιστικές πτυχές και να δίνεται και η κατάλληλη σημασία σε αυτές. Γι' αυτό λοιπόν μην μας λέτε απλώς ότι έχουμε δίκιο και ότι τους φόβους σας τους ημεριζόμαστε, αλλά θέλουμε στο κείμενο ξεκάθαρα να φαίνεται ε, ρητά όλο αυτό που ζητάμε χωρίς να υπάρχουν παρεξηγήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε τέτοιους φόβους γιατί θέλουμε να φροντίσουμε να, για τους ανθρώπους που μας ενδιαφέρουν, για το θέατρο, για το ραδιόφωνο. Όπως είπε και η κυρία Κάμερεβερτ, πρέπει αυτό να αναφέρεται ξεκάθαρο στο κείμενο. Δεν είμαστε φοβετσιάριδες από τη φύση μας. Τον φόβο τον έχουμε αν δεν βλέπουμε αυτά που θέλουμε στο κείμενο. Υπάρχουν πολλές παγίδες και δεν λέμε ότι θέλετε να μας εξαπατήσετε, αλλά καμιά φορά στο τέλος ε, βλέπουμε ότι αυτό που εσείς με καλές προθέσεις θέλατε να μας βεβαιώσετε ότι θα κάνετε, δεν το βλέπουμε στο τέλος. Για το DVD επίσης έγιναν και κάποιες προτάσεις. Ε, τελειώνουμε με αυτό και πάμε στο σημείο 13. Εχθές έγινε η συνάντηση των συντονιστών και σας στείλαμε τις αποφάσεις με email, τις διαβάσατε, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Για τα διάφορα τώρα στο 14 έχει κανείς να πει κάτι. Όχι, πάμε στο σημείο 15. Στις 24-25 Ιανουαρίου θα συναντηθούμε ξανά. Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε τους διερμηνείς και σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και καλό, καλή χρονιά να είναι το 2011. Ευχαριστούμε.